Yeah. Excuse me, I cannot start because there are some members, but not not all. Δεν μπορώ να αρχίσω, μόνο μερικά μέλη είναι εδώ, δεν είναι όλοι. And we cannot change the draft, that's a problem. Και δεν μπορώ να αλλάξω την ημερήσια διάταξη, αυτό είναι το πρόβλημα. Συνάδελφοι, να σας καλημερίσω στην ε, συνεδρίαση της Επιτροπής μας. Να πω ότι έχουν γίνει κάποιες αλλαγές στην ημερήσια διάταξη. Δεν έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα. Καταρχάς, στο σημείο 4 για την έκθεση του κυρίου Μπουτικόφερ δεν χρειάζεται περαιτέρω συζήτηση. Μπορούμε να περάσουμε κατευθείαν στην ψηφοφορία. Άρα το αφαιρούμε το σημείο υπερθμών 4. Τώρα στο 10 το ίντερνετ των πραγμάτων και αυτό θα το αφαιρέσουμε από την ημερήσια διάταξη γιατί δεν είναι εδώ ο εισηγητής. Δεν μπορώ να το αλλάξω, η εισηγητρία δεν είναι εδώ. δεν μπορώ να το αλλάξω μένα, αλλά μπορώ να σας πω ότι δεν με ικανοποιεί ιδιαίτερα να λείπουν οι εισηγητέ σε περίπτωση που υπάρχει ένα θέμα στην ημερήσια διάταξη. Τώρα για το σημείο 12 του κυρίου Τοσνόφσκι ούτε αυτό θα το συζητήσουμε ασφαλώς, αλλά μπορούμε να το ψηφίσουμε κατευθείαν σήμερα για το εισηγητή με ενημέρωσε ότι σε όλα τα θέματα που αφορούν τις τροπολογίες μπορούμε να περάσουμε σε ψηφοφορία. Αν δεν έχετε λοιπόν αντιρρήσεις, έτσι θα εγκρίνουμε την ημερήσια διάταξη και θα περάσουμε έτσι στο σημείο 3 της ημερήσιας διάταξης, μετά τις ανακοινώσεις ε, του Προέδρου. Δεν είχα κάτι να σας ανακοινώσω στο 2. Στο 3 λοιπόν. Ασφάλεια του εφοδιασμού σε φυσικό αέριο. Το έχουμε συζητήσει πολλές φορές το θέμα αυτό. Θα έχουμε μία ανταλλαγή απόψεων για τις τροπολογίες σήμερα όπως θα διαπιστώσετε κι εσείς, είναι μεγάλος ο αριθμός ε, των τροπολογιών και ο κύριος Βιτάλ Κβάντρας θα πάρει πρώτο το λόγο να μας παρουσιάσει το θέμα αυτό και μετά μπορούμε να το συζητήσουμε από τις 10 ξεκινάει η ψηφοφορία σας υπενθυμίζω με τις ηλεκτρονικές σας κάρτες ο κύριος Βιτάλ Κβάντρας Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε εγώ θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους αυτής της Επιτροπής για την δουλειά τους σε αυτό το σχέδιο κανονισμού. Το ενδιαφέρον που έδειξαν αντικατοπτρίζεται από τον αριθμό των τροπολογιών που είναι 500. Πραγματικά υπάρχει αληθινό ενδιαφέρον για αυτή την νομοθεσία. Αυτό το οποίο θέλω εγώ να σας αναφέρω είναι μία πρώτη ανάλυση αυτών των τροπολογιών οι οποίες σε μεγάλο βαθμό συγκλίνουν και ως προς το νόημά τους και ως προς τις προθέσεις τους. Έχω λοιπόν την εντύπωση ότι δεν θα είναι καθόλου δύσκολο να προχωρήσουμε σε συμβιβασμούς. Έχουμε δύο ομάδες τροπολογιών που μπορούμε να διαχωρίσουμε. Μία που θέλει, θέλουν να βελτιώσουν την πρόταση χωρίς ριζικές αλλαγές στο κείμενο και μερικές οι οποίες είναι σαφώς πιο ριζικές και προτείνουν ουσιαστικότερες αλλαγές. Είπαμε λοιπόν υπάρχουν οι βελτιωτικές τροπολογίες χωρίς να αλλάζουν ε, τα πράγματα και να σας αναφέρω τις εξής. Μερικές οι οποίες τονίζουν το ρόλο της αγοράς ως πρώτη φάση πρόληψης της κρίσης. Κανένα πρόβλημα γι' αυτό. Άλλες θέλουν να δώσουν μεγαλύτερη βαρύτητα στην ομάδα συντονισμού φυσικού αερίου, περισσότερη διαβούλευση, περισσότερο συντονισμό. Ούτε και σε αυτό έχουμε πρόβλημα. Επίσης έχουμε τροπολογίες οι οποίες θέλουν να βρουν τον κατάλληλο τρόπο ούτως ώστε το κόστος και οι επένδυσεις στις νέες υποδομές να κατανέμεται ισορροπημένα μεταξύ αυτών που επενδύουν και των δικιούχων. Ούτε και εδώ έχουμε πρόβλημα. Έχουμε επίσης και τροπολογίες οι οποίες αφορούν στην οικονομική αποτελεσματικότητα, στην ασφάλεια του ανεφοδιασμού ε, ως προϋπόθεση ε, για την ε, δημιουργία της υποδομής. Και εδώ συμφωνούμε. Έχουμε και τροπολογίες οι οποίες θέλουν να είμαστε πολύ πιο προσεκτικοί με τις ρήτρες, ρήτρες προορισμού κλπ. όταν συνάπτουμε συμφωνίες με τρίτες χώρες. Και σε αυτό μπορούμε να βρούμε λύσεις. Και μετά έχουμε άλλες που τονίζουν ότι είναι αναγκαίο να έχουμε σύνδεσεις δικτύων για να συνδέσουμε περιοχές οι οποίες είναι ε, κέντρα παραγωγής ενέργειας. Αυτή είναι η πρώτη κατηγορία λοιπόν τροπολογιών. Έχουμε και άλλες οι οποίες τονίζουν ε, τη σημασία των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ε, την ασφάλεια στον ανεφοδιασμό. Όλα αυτά είναι συζητήσιμα χωρίς προβλήματα δεύτερη κατηγορία είναι αυτές ε, που θέλουν πιο ουσιαστικές αλλαγές. Εγώ τις ξεχώρισα στις εξής κατηγορίες. Ο ορισμός προστατευμένου πελάτη. Οι περισσότερες τροπολογίες τίνουν προς την κατεύθυνση ενός ευρωπαϊκού ορισμού για να αποφύγουμε καταχρήσεις για να ανταποκριθούμε σε αυτήν την λογική ανησυχία, εγώ πρότεινα σε ευρωπαϊκό επίπεδο ο ορισμός να περιορίζεται στα νοικοκυριά. Λοιπόν, αυτό κοινό για όλη την Ευρώπη. Τα νοικοκυριά είναι προστατευμένα, διότι το στάνταρ του ανεφοδιασμού συνδέεται με αυτόν τον ορισμό. Τώρα, εάν ένα κράτος μέλος έχει επαρκείς δυνατότητες για να εγγυθεί ασφάλεια και σε άλλους καταναλωτές μπορεί να το κάνει. Φτάνει να μην υποσκάπτει την αλληλεγγύη με τους γειτόνους του σε περίπτωση ανάγκη και χωρίς υποχρέωση για τα άλλα κράτη-μέλη σε περίπτωση κρίσης να καλύπτουν αυτήν την επιπλέον ζήτηση. Έτσι λοιπόν πρόσθεσα μερικά άλλα στοιχεία για την ανάλυση του κινδύνου και τα προληπτικά σχέδια σχετικά με αυτή τη δυνατότητα. Και δεν θα είχα και πρόβλημα να προσθέσω ένα κριτήρια όπως προτείνει ο συνάδελφος Βόμποντα ούτως ώστε αυτοί οι επιπλέον πελάτες να είναι ειδικέ ε, δημόσιες υπηρεσίες. Δεν έχω πρόβλημα λοιπόν. Αλλά άλλοι συνάδελφοι θέλουν να αλλάξουν τις προδιαγραφές του L-1 αντί δηλαδή υποχρεωτική προδιαγραφή να έχουμε δίκτυ. Αυτή είναι μια πολύ δραστική αλλαγή στη φιλοσοφία του κανονισμού. Κατά τη γνώμη μου, το κριτήριο νη μείον ένα πρέπει να είναι δεσμευτικό. Πάντα στο βαθμό που το τελικό παράρτημα θα είναι τεχνικά σωστό, μπορεί να εφαρμοστεί σε τονίζω περιφερειακό επίπεδο και εγκαιάται συγκρίσιμα αποτελέσματα μεταξύ των κρατών μελών. Το N, το νη πρέπει να είναι καρπός της ανάλυσης του κινδύνου, των επιπτώσεων και της δυνατότητας των κρατών μελών να καλύπτουν τις προδιαγραφές λαμβάνοντας υπόψη τις εθνικές ιδιομορφίες. Δεν πρέπει να είναι δηλαδή ένας ε, ε, σιδερένιος ε, κορσές ίδιος για, τους, για όλους. Πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη την ετερογένεια των αγορών φυσικού αερίου στην Ευρώπη. Αλλά το να το υποβαθμίσουμε και να γίνει από υποχρεωτικός όρος απλώς δείκτης ε, δεν γίνεται. Πρέπει να τα βρούμε λοιπόν μεταξύ αυτών των δύο απόψεων. Επίσης είμαι ικανοποιημένο και το λέω εδώ στην Επιτροπή ότι στο Συμβούλιο υπάρχει μία συνένεση για τον ή μείον ένα να είναι υποχρεωτικό. Λοιπόν τώρα άμα το Συμβούλιο δηλαδή θέλει να είναι υποχρεωτικό τον ή μείον ένα, εμείς τώρα γιατί να τα ανακατέψουμε τα πράγματα. Άλλο σημείο προβληματικό είναι το παράρτημα, είναι το τμήμα μάλλον για τη διαχείριση κρίσης. Και εδώ έχουμε τροπολογίες για όλα τα γούστα. 10%, 20%. Ποια θα είναι η αρμόδια αρχή, θα είναι μία αρχή, δύο αρχές, ε, θα, τι θα γίνει, θα, θα, πώς θα ορίζεται, θα έχουμε ε, ε γεωγραφική τοπική, ε, αυτές οι τροπολογίες είναι ενδιαφέρουσες και όλες ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Εμένα όμως η προσωπική μου γνώμη είναι ότι δεν θα πρέπει να περιορίζουμε τη δυνατότητα κήρυξης ε, κοινοτικής έκτακτης ανάγκης. Σίγουρα υπάρχουν εθνικές περιπτώσεις που ορισμένες φορές μπορεί να είναι πολύ σοβαρές ή περιφερειακές. Αλλά μην παρακολύουμε ε, τη δυνατότητα κήρυξης ε, κοινοτικής έκτακτης ανάγκης. Αν κάνουμε εμείς ε, έναν εξαντλητικό κατάλογο των διαφόρων καταστάσεων υποχρεώνοντας την Επιτροπή να κηρύσει η κατάσταση έκτακτης ανάγκης όταν, μια, όταν ένα κράτο το ζητάει, όταν ε, μεσολαβεί κάτι το πολύ σοβαρό σε ένα κράτος μέλος, τότε εμεί κλείνουμε την πόρτα στη δυνατότητα της Κομισιόν να κηρύσει κοινοτική εκτακτη ανάγκη η οποία μπορεί να ευεργετεί τις χώρες που πλήττονται πιο άμεσα. Πρέπει να το έχουμε λοιπόν αυτό ως πιθανότητα. Είναι ένα σημείο πολεμικής αυτό. Εγώ ελπίζω ότι θα μπορέσω να προτείνω έναν συμβιβασμό που θα εγγυάται ότι αν ένα ή πολλά κράτη-μέλη αντιμετωπίζουν κρίση και περιορίζεται σε, αυτή η κρίση είτε σε μια μικρή ομάδα κρατών μελών ή μόνο σε ένα κράτος μέλος, αυτό το κράτος μέλος να μην μένει απροστάτευτο, να τη χάνει της αλληλεγγύης της υπόλοιπης Ένωσης. Θέλω λοιπόν εγώ να πληροφορήσω τους την αναδέλφους ότι η γραμματεία της Επιτροπής σας έστειλε ένα νέο κείμενο που ε, μας ε, έστειλε και το, Συμβούλιο για την Περιφερειακή Συνεργασία πρόκειται για ένα νέο παράρτημα όπου ορίζονται ποιες είναι εκείνες οι περιοχές, οι περιφέρειες της Ένωσης όπου θα πρέπει να υπάρχει συνεργασία για την ασφάλεια στον ανεφοδιασμό. Πολλοί συνάδελφοι της Επιτροπής εκφράστηκαν λέγοντας ότι στο κείμενο θα πρέπει να ενισχύσουμε την περιφερειακή διάσταση την περιφερειακή συνεργασία που είναι ο καλύτερος τρόπος για να ανταποκριθούμε σε μια κρίση ανεφοδιασμού. Εγώ συμφωνώ απόλυτα με αυτήν την τοποθέτηση και είμαι απόλυτα πεπισμένος ότι ένα κομμάτι από το πρόβλημα, ένα τμήμα του προβλήματος που αναφέρω εδώ για την κήρυξη κοινοτικής έκτακτης ανάγκης μπορεί να αντιμετωπιστεί μέσα από μια περιφερειακή εστίαση. Τώρα αγαπητοί συνάδελφοι, κύριε Πρόεδρε, αυτό το κείμενο του Συμβουλίου ε, μας ήρθε εκτός προθεσμίας κατάθεσης τροπολογιών. Και τώρα δεν είναι εύκολο να το εισάγουμε στην ψηφοφορία ή να το συζητήσουμε. Πιστεύω λοιπόν ότι η λύση εναπόκειται στο ότι εγώ ως εισηγητής και, και όλοι οι εισηγητές να επεξεργαστούμε ένα κείμενο του Κοινοβουλίου και αν συμφωνήσουμε να το ψηφίσουμε σε αυτήν την Επιτροπή εάν φυσικά η Προεδρία και οι συντονιστές των ομάδων θεωρούν ότι είναι σωστό. Φυσικά όλα τα μέλη της Επιτροπής μπορούν να στείλουν προτάσεις για να βελτιώσουμε αυτό το κείμενο. Άλλες τροπολογίες οι οποίες αλλάζουν σημαντικά την πρόταση είναι να αυξήσουμε τις εξουσίες της Κομισιόν σε περίοδο κρίσης. Είναι οι τροπολογίες εκείνες που δίνουν την δυνατότητα να παρεμβαίνει η Κομισιόν άμεσα στην αγορά άμα δεν ικανοποιείται από τη δράση των κρατών μελών. Εγώ όμως έχω αμφιβολίες ότι κάτι τέτοιο είναι πολιτικά εφικτό. Είναι φυσικά λογικό να ακούσουμε την Κομισιόν που είναι και ο άμεσα ενδιαφερόμενος και η Κομισιόν να εκφραστεί σχετικά. Εγώ πάντοτε ήμουνα υπέρ του η Κομισιόν να έχει μία σειρά δυνατοτήτων και αρμοδιοτήτων ώστε να διασφαλίζει την εύρυθμη λειτουργία όλου του συστήματος σε περίοδο κρίσης ανεφοδιασμού. διότι πολλά κράτη-μέλη δεν θα το δεχθούν η Κομισιόν να έχει σε τέτοιου είδους περιστάσεις απόλυτη εξουσία. Θα προσπαθήσουμε λοιπόν να βρούμε και εδώ μία λογική σύγκληση. Υπάρχουν επίσης και τροπολογίες οι οποίες ζητούν περισσότερη προσοχή για την εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, η ρήτρα τρίτων χωρών, ελεύθερη κυκλοφορία φυσικού αερίου, ε, ανάπτυξη ενός μηχανισμού έγκαιρης προειδοποίησης. Αυτά είναι πολύ λογικά, μπορούμε κάλλιστα να τα συμπεριλάβουμε στην έκθεση. Και συμφωνώ επίσης και με τις τροπολογίες εκείνες που λένε συνεργασία μεταξύ του κυρίου Έτιγκερ, δηλαδή του Επιτρόπου για την Ενέργεια και της κυρίας Άστον. Αλλά και εδώ προσοχή, διότι αυτή η συνεργασία θα πρέπει να είναι ναι μεν στενή, αλλά και ισορροπημένη, διότι οι συνάδελφοι των εξωτερικών υποθέσεων ε, υπερτιμούν ε, αρκετά το ρόλο της ε, ΥΠΑ του αρμόστρια σε περίοδο ε, ενεργειακής κρίσης. Ξέρετε ότι μία ενεργειακή κρίση ε, κρύβει και πάρα πολλές τεχνικές πλευρές. Σύμφωνη συνεργασία, αλλά ισορροπημένη συνεργασία. Και τελευταίο, πολλά μέλη προτείνουν αρμόδια αρχή να είναι οι εθνικοί ρυθμιστές. Εγώ δεν λέω να αυτό κακή ιδέα. Αλλά μία πλειοψηφία στο Συμβούλιο θα φέρει αντιρρήσεις. Στο τελικό κείμενο πρέπει να λέμε αν η αρμόδια αρχή δεν είναι ο ρυθμιστής, στην προκειμένη περίπτωση δηλαδή η κυβέρνηση, οι δύο αρχές, δηλαδή η εκτελεστική και ο ρυθμιστής, να μπορούν να συνεργάζονται. Πάλι λοιπόν εδώ αναζήτηση της ισορροπίας. Σε γενικές γραμμές αυτή ήταν η περίληψη των τροπολογιών, του περιεχομένου τους, της γενικής αντίληψης που η κάθε μια από αυτές θέλει να εισάγει στην έκθεση και από τώρα και στο εξή, από τώρα και μετά μάλλον, ε, σε συνεργασία με όλους τους ε, συναδέλφους ε, και υπό το όμα των συντονιστών θα ψάξουμε τους συμβιβασμούς. Θα αναζητήσουμε να βρούμε συμβιβασμό, καλό συμβιβασμό σε όλα όσα είπα. Καλή θέληση χρειάζεται και συνεργασία, επικοδομητική συνεργασία. Υπάρχουν πολλές προσδοκίες σχετικά με αυτόν τον κανονισμό. οι ενδιαφερόμενοι φορείς αλλά και η ευρωπαϊκή κοινωνία. Να κοιτάξτε τον τύπο των προηγουμένων εβδομάδων. Ε, τρέφουν πολλές προσδοκίες για αυτόν τον κανονισμό και εμείς ως Επιτροπή δεν πρέπει να τους διαψεύσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πολύ και εγώ. Ευχαριστώ τους συναδέλφους. Για την παρουσίαση αυτή. Έχουμε ακόμα μισή ώρα στη διάθεσή μας και μετά θα πρέπει να διακόψουμε γιατί θα ακολουθήσει η ψηφοφορία. Έξι άτομα έχουν ζητήσει το λόγο. Επτά μάλλον. Αυτό όμως δεν θα, θα κλείσει το κατάλογο των ε, ομιλητών. Και μετά θα θέλαμε να ακούσουμε και τον ομιλητή και τον εισηγητή και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο κύριος Βόμποντα, καταρχάς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω τον συνάδελφο Βίδαλ Κουάτρας. Αν με ακούσει βέβαια και με τον ενοχλούν άλλοι διάφοροι. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον συνάδελφο Βιντάλ Κουάτρας για την ε, δουλειά του είναι πραγματικά δύσκολος ο δρόμος που θα πρέπει να βρούμε, αλλά θα είμαστε σε θέση, ελπίζω, να τον βοηθήσουμε για να φτάσει στο Σαντιάγκο, για να ανοίξει τον δρόμο. Να μιλήσουμε για τα αμφιλεγόμενα. Δεν υπάρχει λόγος να συζητήσουμε θέματα τα οποία δεν παρουσιάζουν πρόβλημα. Καταρχάς, ότι αφορά τα ε, προστατευόμενα εδάφη. Νομίζω ότι θα πρέπει να προσθεθεί στο τοπόθεμα στον προπολογισμό και να μην είμαστε αντίθετοι στην αρχή της ε, επικουρικότητας. Συμφωνούμε απόλυτα. Έχουν γίνει διάφορες ε, προτάσεις και από το, την ομάδα μου. Εγώ πιστεύω ότι, συνάδελφε, θα πρέπει να μείνουμε στα υποχρεωτικά επίπεδα αν θέλουμε να υπάρχει κάποια ευελιξία στις εθνικές κυβερνήσεις. Αν αρχίσουμε να μιλάμε τώρα ήδη για δείκτες και μετά κάνουμε προσαρμογές, ε, θα ήταν πιο δύσκολα τα πράγματα. Σας στηρίζω λοιπόν. Σε ό,τι αφορά θέματα κρίσης, νομίζω ότι ελπίζουμε να μην τεθεί σε εφαρμογή η νομοθεσία αυτή, γιατί ελπίζουμε να μην χρειαστεί να μην παρουσιαστεί τέτοια κρίση. Αλλά αν παρουσιαστεί τέτοια κρίση, ελπίζω να μπορέσει να ανταποκριθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ε, περιφερειακή συνεργασία. Μου αρέσει η πρόταση της, ε, του εισηγητή, αλλά μου κάνει εντύπωση ότι στον κατάλογο των χωρών που πλήττονται αναφέρεται και η Σλοβακία. Γιατί δεν ε, περιλαμβάνεται η Σλοβακία σε κάποια περιφερειακή ένωση. Δηλαδή η Σλοβενία περιλαμβάνεται, η Ουγγαρία περιλαμβάνεται, αλλά όχι η Σλοβακία. Αυτό είναι λεπτομέρεια και σε ό,τι αφορά τις δυνατότητες αγοράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αν θέλουμε ε, να ορίσουμε το πλαίσιο της δυνατότητας παρέμβασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αν θέλουμε λοιπόν και ορίσουμε με σαφέ τρόπο το πλαίσιο μας το οποίο μπορεί να επέμβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ε, δεν θα έχουμε πρόβλημα. Δηλαδή, θα μπορούμε να ορίσουμε ότι καταρχά αρμόδιε οι οι εθνικέ αρχέ και μετά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Φυσικά θα μπορούν να γίνουν προσαρμογέ, αλλά αν υπάρχει μια γενική αρχή. Τώρα η συνεργασία Ουτίνγκερ Άστον. Και αυτό είναι ένα θέμα ε, το οποίο θα πρέπει να το δούμε στην πράξη. Δεν βλέπω να υπάρχει κάποια αντίπαλότητα μεταξύ των δύο θέσεων. Από εκείνου θα πρέπει να δράσουν αυτοί οι δύο σε διπλωματικό επίπεδο δηλαδή Άστον, σε πιο ε, τεχνικό επίπεδο ο κύριος Έτινγκερ σε ό,τι αφορά τις επαφές για παράδειγμα με τους, ε, τις εταιρείες ε, δεν βλέπω να υπάρχει κάποια αντίφαση και θεωρώ ότι υπάρχει ε, μεγάλο περιθώριο για <coughs> συμβιβασμούς. Για να μπορεί να αντιδρά γρήγορα το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Δεν θέλουμε να βάλουμε φραγμού σε οτιδήποτε, να βάλουμε εμπόδια. Νομίζω ότι είναι, θα είναι ένα καλό μήνυμα αυτό από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, να προωθηθεί δηλαδή γρήγορα το θέμα. Ευχαριστώ κύριε Τσιμάνσκι. Ε, λοιπόν, χωρί μικρόφωνο ο μιλητής. Ήθελα λοιπόν να σας πω ότι πραγματικά ευγνωμονώ και συγχαίρω τον εισηγητή διότι θα μας βοηθάει να λύσουμε το πρόβλημα των 500 τροπολογιών και να τελειώνουμε με αυτόν τον κανονισμό ο οποίος τελικά πληρεί τις αρχές της Λισαβόνας ε, για την αλληλεγγύη μεταξύ των χωρών. Ε, παίζονται πάρα πολλά πράγματα κύριε Βίδαλ Κουάδρας με αυτόν τον κανονισμό. Αν εμείς θέλουμε ένα μέσο το οποίο πραγματικά να έχει επιπτώσει στη βελτίωση της ασφάλειας του ανεφοδιασμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει να έχουμε σαφώς ορισμένο τον ρόλο της Κομισιόν, πώς παρεμβαίνει δηλαδή στην αγορά και με τη μέσα. Πραγματικά συγχαίρω απόλυτα την ε, συντονιστική ομάδα. Ε, πίστευω ότι πρέπει να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι όλα αυτά μπορεί να είναι ανεπαρκή σε περίπτωση σοβαρής κρίσης. Και ο ρόλος της Κομισιόν στην προκειμένη περίπτωση είναι πάρα πολύ σημαντικός. Και αυτό το 10% προς μία χώρα είναι κάτι το πάρα πολύ σημαντικό, διότι αλλιώ θα καταλήξουμε σε έναν κανονισμό που δεν θα λειτουργήσει ποτέ. Και μπορεί να δημιουργήσει δυσχέρειες και για τα κράτη-μέλη και για τους πολίτες που θα πληρώσουν την ύφη το θέμα των προστατευμένων καταναλωτών. Μα και αυτός και, ο τομέας δεν μπορεί να είναι ιδιαίτερα ευρύς, ε, διότι σε περίπτωση κρίσης πρέπει να είμαστε σαφείς, να στοχεύουμε σε κάτι. Και επίση για τις επενδύσεις χρειαζόμαστε τεράστιες επενδύσεις στον τομέα των υποδομών, στην σύνδεση, στα διαδίκτυα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό λοιπόν κύριε Σιγητά θα πρέπει να εργαστούμε σοβαρά γύρω από τους μηχανισμούς αντιστάθμισης του κόστους των επενδύσεων. Δεν μπορούμε όμως να υποστηρίζουμε τις τροπολογίες οι οποίες αντίκυνται σε αυτού του είδους τις επενδύσεις, διότι αυτές οι επενδύσεις είναι πάρα πολύ σημαντικές για να μπορέσουμε να ε, καταλήξουμε στην πολιτική των υποδομών. Συμφωνώ με τον κύριο Ζάριους Βόλσκι, είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα των τροπολογιών ε, για την συνεργασία με την κυρία Άστον. Συμφωνώ λοιπόν με τον κύριο Σάριους Βόλσκι, ξαναλέω. Εμείς με αυτόν τον κανονισμό κάνουμε ένα πολύ σημαντικό βήμα στην ασφάλεια του ενεργειακού ανεφοδιασμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εμείς ε, δίνουμε ένα σημαντικό μέσο στα χέρια των πολιτών. Βλέπουν η διεισόμαση ότι η Ένωση αλλάζει μετά από τη συνθήκη της Λισαβόνας και έχουμε πραγματικά προστιθέμενη αξία. Σας ευχαριστώ λοιπόν κύριε Βιδάλ Κουάδρας για τη δουλειά που κάνατε. Ε, Ο κύριος Τούρμης, ευχαριστώ. Καταρχάς ε, να πω ότι Αλέχο, έχεις αναλύσει σωστά την κατάσταση και τώρα θα πρέπει να ψηφίσουμε πλέον. Θα πρέπει να ψηφίσουμε όχι μόνο ακολουθώντας μια καλή φιλοσοφία σε θέματα όπως ε, την πρόληψη των κρίσεων και την εισαγωγή μέτρων, τον καλό συμψηφισμό, αν θέλετε, ισορροπία μεταξύ ε, Αγορά και ασφάλεια και ύστερα το επίπεδο το τοπικό, το περιφερειακό και το επίπεδο τη Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Όλα αυτά θα πρέπει να τα ψηφίσουμε, αλλά θα πρέπει να ψηφίσουμε σε ό,τι αφορά κάποια στοιχεία αναφορικά με το Συμβούλιο. Συνάδελφε, λοιπόν, θα πρέπει να δείξουμε στρατηγικό πνεύμα κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας. Έχω υποβάλει ε, τροπολογίες για τις ε, αναδρομικές ροές Πολύ σημαντικό αυτό, είναι φτηνό και θα αποφέρει πολλά. Ένα άλλο θέμα είναι όσο πιο πολύ εξουσία γίνεται στις ρυθμιστικές υπηρεσίες. Θεωρώ ότι υπάρχει μεγάλος κίνδυνος αν οι ρυθμιστικές αυτές υπηρεσίες δεν είναι αυτές που θα καθοδηγούν το σύστημα, γιατί θα έχουμε στα περίπτωση αυτή δύο εθνικές αρχές που θα ανταγωνίζονται η μία την άλλη και θα πρέπει να υπάρχει μια υψηλότερη αρχή η οποία θα υποσκάπτει αν θέλετε την εξουσία των ε, υπηρεσιών αυτών. Χρειαζόμαστε λοιπόν τέτοιες υπηρεσίες οι οποίες θα είναι στη θέση του οδηγού και θα πρέπει επίσης να αυξηθεί και η διαφάνεια. Ένα βασικό θέμα θα αποτελέσει και η όσο πιο περιοριστική ερμηνεία είναι δυνατόν της προστασίας των πελατών. Και διάβασα και τις ε, τροπολογίες της κυρίας Νίμπλερ και του καθεξής. Νομίζω ότι αυτή τη γραμμή θα πρέπει να ακολουθήσουμε. Δεν πιστεύω ότι ο προπολογισμό της Ένωσης θα μας βοηθήσει να επιλύσουμε το θέμα των επενδύσεων στο φυσικό αέριο. Νομίζω, συνάδελφοι, δεν πρόκειται να έχουμε δισεκατομμύρια στη διάθεσή μα ε, από τον προπολογισμό της Ένωσης. Αυτό που θα κάνουμε με την οδηγία αυτή είναι να ρυθμίσουμε την κατάσταση, να βρούμε ένα σύστημα ρύθμισης το οποίο θα υποχρεώνει τους φορείς να λαμβάνουν μέτρα προληπτικά, αν θέλετε, όπως αυτό της ε, αναδρομικής ροής. Και πολύ φοβάμαι ότι ούτε ΝΑΙ, ούτε η Eurocas, ούτε ο ΣΟΕΣ δεν είναι φτωχέ αυτές οι εταιρείε. Έχουν πολλά χρήματα όλοι αυτοί. Αλλά θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι τα χρήματα αυτά θα κινηθούν προς τις σωστές επενδύσεις. Γι' αυτό χρειαζόμαστε τις, ε, τη ρύθμιση. Δεν είναι ο Άι Βασίλης ε, το Ευρωπαϊκό προπολογισμό. Χρειαζόμαστε σκληρή ρύθμιση. Δύο ερωτήσει να κάνω προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Καταρχάς σε ό,τι αφορά αυτό το ε, περιφερειακό επίπεδο. Και εγώ, και εγώ το επιθυμώ αυτό, αλλά πολύ φοβάμαι ότι αν δεν επιδείξουμε την απαραίτητη προσοχή θα περάσουμε σε περιφερειακό επίπεδο με λιγότερε όμω υποχρεώσει σε ό,τι αφορά τι λεπτομέρειε. Και εσείς ερμηνεύοντας το κείμενο του Συμβουλίου είστε σίγουροι ότι δεν υπάρχουν παραθυράκια. Μήπως κάτι θα πρέπει να διορθώσουμε. Και ένα τελευταίο θέμα που με απασχολεί ιδιαίτερα. Α, με ανησύχησε ιδιαίτερα αυτό που συνέβη στην Πολωνία. Δηλαδή έξι μέρες την εβδομάδα α, έχουμε θέματα ανταγωνισμού, μετά έχουμε θέματα με τη Ρωσία και την τελευταία ημέρα έχουμε μελέτη για την Gazprom. Δηλαδή τι, αποδεχόμαστε και μία ρήτρα προορισμού η οποία είναι κατά του ανταγωνισμού. Αυτό θα είναι, αυτή θα είναι η κατάσταση. Το επιχείρημα δηλαδή της ασφάλειας ανεφοδιασμού θα υποσκάψουμε την ε, ενιαία αγορά. Τι σκοπεύει να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως προς αυτό. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος, ο συνάδελφος Βαλέαν. Η κυρία Βαλέαν. Εκτός μικροφώνου. Micro, First, thank you. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Βιδάλ Κουάντρας για την εξαιρετική αυτή δουλειά για πολύ δύσκολα θέματα. Θα ήθελα να απευθυνθώ να, να αναφερθώ σε κάποια από αυτά. Καταρχάς για τον μείον 1. Αρχικά θεωρούσα ότι δεν θα έπρεπε να χρησιμοποιηθεί ως πρότυπο αλλά ως ε, δείκτης πιο πολύ. Και με ανησύχησε γιατί μπορεί να αποτύπωνε με στρεβλωμένο τρόπο αυτό το αίσθημα της ε, ασφάλειας και αν θέλετε θα άφηνε μεγάλο περιθώριο ερμηνεία. Ωστόσο τώρα πλέον τίμουν να πιστέψω ότι αυτό το μέσο παρά το ότι δεν θα είναι τέλειο, καλό θα είναι να ορίσει ένα ελάχιστο κατόφλι. Δεσμευτικό. Ιδάλλως μπορεί να μην έχει αποτέλεσμα καθόλου αυτή η οδηγία. Φυσικά θα πρέπει να προσέξουμε κατά την εφαρμογή του μέσου αυτού και να λάβουμε υπόψη και τις τοπικές, ε, τις ανάγκες του κάθε, καθούς, του κάθε κράτους μέλους βλέπουμε ότι με την νομοθεσία αυτή δίνεται σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ευρείες αρμοδιότητες στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και εγώ συνήθω δεν είμαι υπέρ της αρχής αυτής. Καταλαβαίνω ότι θα είναι κρίσιμο ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά το συντονισμό τέτοιων σχεδίων έκτακτης ανάγκης. Δεν θα πρέπει να έχει τόσο μεγάλη δυνατότητα προσαρμογής μας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να είναι μια πρόσθετη αξία, αν θέλετε. να μην επεκταθούν περαιτέρω σε καμία περίπτωση οι αρμοδιότητές της. Γι' αυτό λοιπόν καλωσορίζω τον ε, μεγαλύτερο ρόλο του Συμβουλίου για την ε, πρόληψη, για τον συντονισμό του αερίου, αλλά μέχρι εκεί. Για την περιφερειακή συνεργασία πιστεύω ότι η πρόταση του Συμβουλίου η οποία μας μεταφέρθηκε, μας διαβιβέστηκε, είναι ενδιαφέρουσα και θα πρέπει να λάβουμε υπόψη το παράρτημα υπαριθμών 4 γιατί ενισχύει την περιφερειακή συνεργασία όταν μιλάμε για την ασφάλεια του εφοδιασμού και υπό την έννοια αυτή θα ήθελα να επιμείνω σε μια πιο μακροπρόθεσμη προοπτική. Θα πρέπει θεωρώ να υπάρχουν εναλλακτικές ε, πηγές και οδοί εφοδιασμού. Τέλος, για το κατόφλι. Τέλος για κήρυξη ε, κατάστασης εκτάκτου ανάγκης. Δεν νομίζω ότι υπάρχει ε, λόγος να θεθεί ένας αριθμητικός, ένα αριθμητικό στοιχείο. Θεωρώ ότι έχουμε ακόμα κάποια δουλειά να κάνουμε για να βρούμε μια σωστή λύση για το πρόβλημα αυτό και το χειρότερο σενάριο θα ήταν ε, να είναι τόσο τελικά περιοριστική και αυστηρή αυτή η νομοθεσία, αυτή η οδηγία που τελικά τα κράτη-μέλη μπορεί να περάσουν μια κρίση χωρίς να έχουν τη δυνατότητα να επικαλυστούν το μέσο αυτό, γιατί τους υπολείπεται για παράδειγμα 1%. Θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο το σύστημα αυτό να ανταποκρίνεται σε όλες τις ε, ενδεχόμενες καταστάσεις, τηρώντας τις αρχές της επικουρικότητας. Ε, και ανυπομονώ να συζητήσω το θέμα αυτό και με τον κύριο Κουάτρας, αλλά και με τους Κιώτης. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Να παρακαλέσω τους επόμενους ε, ομιλητές να τηρήσουν το χρόνο τους, παρακαλώ. Ε, Πρόεδρε, ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστώ θερμά τον συνάδελφο Βιτάλ Κουάντρας, ο οποίος συνέβαλε τα μάλα στη δουλειά αυτή. Είμαι πεπισμένος ότι η υποστολή μας θα ολοκληρωθεί επιτυχώς. Και μάλιστα είναι αυτό το χρόνο όταν έχουμε τον κανονισμό ε, την ώρα που χρειάζεται, δηλαδή να είναι έτοιμος την ώρα που χτυπάει η κρίση, που ενσκύπτει η κρίση. Που εγκύπτει η κρίση. Ε, δεν μπορώ όμως να μπω σε όλες τις λεπτομέρειες του θέματος, διότι Εάν πρέπει να εξασφαλίσουμε αποτελεσματική λειτουργία κάθε στοιχείου του δικτύου προμήθειας αερίου θα πρέπει κάθε χώρα να είναι συνδεδεμένη σε ένα δίκτυο ευρωπαϊκό, σε ένα δίκτυο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πράγμα το οποίο όμως δεν ε, επιλύει το πρόβλημα των ενεργειακών νήσων Εχθές έθεσα και το ερώτημα του πώς μπορεί να επιληθεί το πρόβλημα των ενεργειακών νήσων και μου δόθηκε απάντηση ότι για τα βαλτικά κράτη θα ληφθεί υπόψη ιδιαιτέρως αυτή η κατάσταση, η ιδιαιτερότητά τους. Τώρα όμως βλέπω ότι για την Ετωνία δεν υπάρχει αυτή η ε, δυνατότητα να τηρήσουμε τον νήμιον ένα. Τώρα μα είπανε ότι μπορεί και να συνδεθούμε με τα δίκτυα. Αλλά το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι και να τηρήσουμε τον ήμιον 1, πάλι είμαστε ενεργειακή νήσος. Δεν είναι βιώσιμη για την Ευρώπη μια κατάσταση κατά την οποία ε, χώρες ολόκληρες, αγορές ολόκληρες θα εξαρτώνται από έναν προμηθευτή για το φυσικό του αέριο, την Gazprom πάνω απ' όλα δεν μπορεί να εξαρτώμεθα από την Gazprom και τους εκβιασμούς της. Όταν υπάρχει ε, ένας ε, προμηθευτής φυσικά ο δρόμος ανοίγει στην κατάχρηση και την ε, και τους εκβιασμούς. Αυτό το έχω δει εγώ στη χώρα μου σε μεγάλο βαθμό. Και βλέπω ότι για το συγκεκριμένο αυτοκανονισμό θα πρέπει να αναλάβουμε συγκεκριμένα μέτρα. Ιδάλλως δεν θα αξίζει ούτε καν το όνομά του αυτός ο κανονισμός για την διασφάλιση των προμηθειών φυσικού αερίου. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση της, ε, ε, να αναλάβει τα κατάλληλα μέτρα, να ε, προσφέρει τους κατάλληλους πόρους ώστε να επιλύσει το πρόβλημα των ενεργειακών νήσων. Σας ευχαριστώ πολύ. Έχουμε ακόμα την Επιτροπή και τον εισηγητή. Και, το, και βέβαια πρέπει να κλείσουμε και για τις ψηφοφορίες τη συζήτηση στις 10 η ώρα. Κύριε Τιτσάου. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Και εγώ θέλω να ευχαριστώ τον κύριο Βιδαλκουάδρας και να υπογραμμίσω πολύ σημαντικά στοιχεία. Είναι καταρχάς πολύ σημαντικό για τους ε, ε, προστατευόμενους καταναλωτές, να εξασφαλίσουμε τους θεσμούς που θα προσφέρουν ε, την ε, υπηρεσία όπως αυτή χρειάζεται, όπως επί παραδείγματι οι μονάδες προσφέρουν τα βασικά τρόφιμα στον καταναλωτή. Το ίδιο θα πρέπει να υπογραμμίσουμε την έννοια της αλληλεγγύης, κοινωτικής αλληλεγγύης σε περιόδους ενεργειακής κρίσης και ελπίζω στην έκθεση κ. Βαλίαν να γίνουν ε, δεκτές οι τροπολογίες οι οποίες ε, ε, βάλουν κατά του κατακαιρματισμού, δηλαδή εκείνες οι οποίες εντοπίζουν τις ενεργειακές νήσους. Και επίσης προτείνουν την ενίσχυση των δεσμών με επενδύσει των δεσμών μετά των νήσων αυτών. Γιατί αναφέρομαι στην έκθεση Βαλιάν, διότι, στην τροπολογία συγγνώμη, Βαλιάν, διότι αναφέρεται γενικά στι ενεργειακέ υποδομές και όχι μόνο το φυσικό αέριο πρώτον και δεύτερον διότι θα πρέπει να εισαχθούν οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και να εντοπιστούν οι πηγές ανεφοδιασμού. Ε, σχέδια όπως το Ναμπούκο θα έπρεπε εν προκειμένου να ενσωματωθούν στο καθεστώς Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τον κανονισμό για την διασφάλιση των προμηθειών σε φυσικό αέριο και ιδιαίτερα για να αποφεύγουμε τις ε, ελλείψεις φυσικό, σε φυσικό αέριο. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Νίμπλερ έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Και πολύ σύντομα ευχαριστώ τον εισηγητή μας, τον Αλέχο Βιδαλκουάτρας έδωσε με πολύ αλθρωμένο τρόπο στην εισήγησή του τα βασικά στοιχεία της συζήτησης σήμερα το πρωί. Τρία είναι τα σημεία που θεωρώ πιο σημαντικά. Καταρχάς, τον ορισμό του, της ομάδας των προστατευόμενων καταναλωτών και ευχαριστώ πολύ τον Κλωτ Τσουρμές για τη στάση του που είναι σπάνιο να παρουσιάζει κενό κάποια δική τοποθέτηση αλλά ασφαλώς τον ευχαριστώ πολύ για την ε, επισήμανση και θα υποστηρίξουμε τις προτάσεις εδώ στην Επιτροπή. Δεύτερον, για την ανάστροφη ροή, reverse flow, η υποχρεωτική ο υποχρεωτικό προσδιορισμό του reverse flow μέσα σε τρία χρόνια για όλε τι δομέ είναι ίσω υπερβολικά φιλόδοξο. Βεβαίω και θέλουμε να έχουμε τους, ε, ε, τα σημεία διασύνδεση, τα interconnectors, αλλά δεν νομίζω ότι μπορούμε να φτάσουμε σε πέντε χρόνια σε αυτό. Και αυτό θα ήθελα να υποστήριξω στις τροπολογίες 265 και 266. Και για τον κύριο Ρούμπιχ θα έλεγα ότι θα πρέπει να αποφεύγουμε τις τρευλώσεις της αγοράς και μπορούμε ή πρέπει να ε, θεσπίσουμε ένα σύστημα το οποίο σε τρία στάδια θα μας ε, απαλλάσσει από τις ε, δυσκολίες, από τα προβλήματα. Και επίσης για τους ε, συναδέλφους για να κλείσω θα ήθελα να σημειώσω ότι πιστεύω πως θα πρέπει στον κανονισμό αυτό να προσδιοριστεί ξεκάθαρα το πεδίο των ευθυνών και των ε, αρμοδιοτήτων των εμπλεκομένων, δηλαδή τι πρέπει να κάνουν τα κράτη-μέλη, τι πρέπει να κάνει η Ευρωπαϊκή Διάσταση, τι πρέπει να κάνουν οι επιχειρήσεις και θα συμφωνήσω με την κυρία Βάλιαν ότι θα πρέπει να ε, εμπλακεί εδώ δραστήρια και η σχετική διεύθυνση. Και βέβαια από την Επιτροπή περιμένουμε συγκεκριμένε προτάσει και δεσμεύσει. Και βεβαίω θα αξιολογήσουμε αναλόγω τι τροπολογίε. Ευχαριστώ κύριο Ράνστορφ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Το μικρόφωνο του μίλητη είναι κλειστό. Τώρα δουλεύει. Είμαι ε, κατά της κατάχρησης του όρου φιλοσοφία και φιλοσοφικός γιατί μας οδηγεί σε γελία ε, συμπεράσματα. Να σας δώσω ένα παράδειγμα σε ένα πρόσφατο ταξίδι μου στην, ε, στις Βρυξέλλες, οδικό. Σταμάτησα ε, στο βενζινάδικο εκεί που κάνουμε το διάλειμμα τέλο πάντων και στις τουαλέτες έγραφε ε, χώρος αναψυχής και φιλοσοφίας. Παρακαλώ να μην καταχρώμεθα αυτών των όρων επιπτέλους. Θα ήθελα εδώ να σημειώσω ότι καταγράφεται η διαβούλευση με τον συγητή στις προτάσεις που βλέπουμε και υπάρχουν κάποια σημεία που θεωρώ πάρα πολύ σημαντικά. Καταρχάς, οικονομική διπλωματία. Λαμβάνουμε υπόψη ότι λόγω της κρίσεως οι πωλήσει της Gazprom έπεσαν κατά 30%, πράγμα το οποίο μεταβάλλει τις συνθήκες και προσφέρει σε εμά στην Ευρωπαϊκή Ένωση δηλαδή αγαστές συνθήκες για οικονομική διπλωματία για να αποφεύγουμε τις ε, τρευλώσεις και τις ε, διακοπές που είδαμε πέρυσι κυρίως. Ε, δεύτερη παρατήρηση, η συμπεριφορά των τραπεζών και κατά τη διάρκεια του ακρό, της ακρόασης του κυρίου Έτσιγκερ επεσήμανα τη διάσταση αυτή και πρέπει να υπογραμμίσω και πάλι το γεγονός ότι οι Τράπεζε δεν υποστηρίζουν πολλά από τα δημοσιονομικά μέσα τα οποία είναι απαραίτητα στην πράξη για την λειτουργία των επιχειρήσεων που ε, συναλλάσσονται σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο. Δεν τηρούν δηλαδή το MT 7799 και σχετικούς όρους που απαιτεί η ε, ρωσική πλευρά. Τρίτη παρατήρηση, θα πρέπει να υποστηρίξουμε την διασυνδεσιμότητα, interconnectivity, κυρίως για να αποφύγουμε τις ε, διακοπές στις προμήθειες. Υπήρξε η δυνατότητα στο παρελθόν να έχουμε διασύνδεση και προμήθεια από τη Λευκορωσία, αλλά δεν ήταν έτοιμα για τέτοιου είδους ε, μεταστροφή τα δίκτυά μας. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντική η διαλειτουργικότητα. Και τέταρτο σημείο, η ανάγκη να ε, δημιουργήσουμε δυνατότητες, δυναμικό αποθήκευσης φυσικού αερίου. Όλα τα άλλα μπορούμε να τα έχουμε, αλλά πρέπει και να ε, βελτιώσουμε αυτή τη διάσταση και πάνω απ' όλα να αξιοποιήσουμε τη διπλωματία του λόγου. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Σκάρετς. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Όπως είπε ο κύριος Κουάδρας, η λειτουργία της εσωτερικής αγοράς αποτελεί ασφαλώς μία από τις κύριες εγγυήσεις της απρόσκοπτης προμήθειας ε, φυσικό αέριο, αλλά υπόθηκε ήδη και από άλλους συναδέλφους ότι θα πρέπει να υπάρξει η αλληλοσυνδεσιμότητα. Εάν δεν μπορούμε να έχουμε το προϊόν στη θέση μας, θα πρέπει να μπορούμε να το φέρουμε από κάποια άλλη αγορά. Και σε σχέση με τα όσα είπε ο κύριος Τούρμες, πως κατά πάσα πιθανότητα οι επενδύσεις αυτές δεν θα αντιληθούν από τον Ευρωπαϊκό Προπολογισμό αλλά θα χορηγηθούν από τις ε, επιχειρήσεις φυσικού αερίου. Θα ήθελα να επενθυμίσω ότι υπάρχει περίπτωση στη βορειοδυτική Ευρώπη, τις βαλτικές χώρες δηλαδή, όπου οι επιχειρήσεις φυσικού αερίου δήλωσαν ότι δεν πρόκειται να χρηματοδοτήσουν τέτοιου είδους ε, συστήματα διότι είναι μικρή αγορά, ενώ από την άλλη η Gazprom έχει τέτοια δύναμη που μπορεί και τώρα αλλά και για το μέλλον μακροπρόθεσμα να ε, αποτρέπει και να σιγάσει κάθε ανταγωνιστική προσπάθεια. Έτσι λοιπόν για το φυσικό αέριο θα πρέπει να αναγνωρίσουμε την ανάγκη για κάποιο είδους επιδότηση. Δεν μπορεί η αγορά να χειριστεί το ζήτημα αυτό με συνθήκες ανταγωνισμού ε, και να εξασφαλίσει την αλληλοσυνδεσιμότητα ε, Φερρυπίν μεταξύ Λιθουανίας και Πολωνία. γιατί κανεί δεν ήταν διατεθειμένο να το κάνει αυτό. Α αναλογιστούμε λοιπόν πώ μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα, πώ μπορούμε να το λύσουμε με την αρχή τη αλληλεγγύη, με την ενίσχυση τη εξωτερική αγορά. Χρειαζόμαστε την αλληλοσυνδεσιμότητα, χρειαζόμαστε όμω και η δράση τη Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να καταστήσουμε δυνατή αυτή την αλληλοσυνδεσιμότητα. Ευχαριστώ. Έχουμε πολύ λίγο χρόνο τώρα. Η Επιτροπή παρακαλώ μπορεί να δώσει σύντομες απαντήσεις στις ερωτήσεις που διατυπώθηκαν. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε, θα είμαστε δυνατόν πιο σύντομο. Θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστώ τον κύριο Βιδάλ Κουάντρας και ε, τους ε, βουλευτές που έλαβαν το λόγο. Ε, βλέπετε ότι σιγά σιγά προσδιορίζουμε το στόχο μας με πιο συγκεκριμένου όρους και ε, είναι όλο και λιγότερα τα προβλήματα. Χωρί να, να επισέρχομαι στι ε, επιμέρου ε, τροπολογίε, θα ήθελα να υπογραμμίσω ορισμένα σημεία που θεωρώ πολύ σημαντικά. Συμφωνούμε ιδιαίτερω με τον κύριο Βιδάλ Κουάδρα, αλλά και με τα όσα είπαν κάποιοι άλλοι, ο κύριο Σφόμποντα, ο κύριο Τούρμα, η κυρία Νίμπλερ ιδιαίτερω, ότι το πεδίο του προστατευόμενου καταναλωτή θα πρέπει, η πελάτη θα πρέπει να προσδιοριστεί πιο συγκεκριμένα, έτσι ώστε να είναι και πιο ευρεία βεβαίω και ευέλικτη η ευέλικτος ο ορισμός αυτός, αλλά όσο πιο ευέλικτος ε, γίνει τόσο και πιο ασαφής τελικά και γι' αυτό πρέπει να είμαστε κάπως πιο συγκεκριμένοι. Στο 1-1 θα πρέπει να είναι υποχρεωτική η τήρηση του όρου αυτού Μόνο αυτό μπορεί να δώσει αποτελέσματα. Εξήγησε ο κύριο Σαντάκα και κάποιοι άλλοι βουλευτέ ότι για ορισμένα βαλτικά, για τα βαλτικά κράτη κυρίω και, και άλλα κράτη, ίσω να μην μπορεί να τηρηθεί ο όρο του νήμιον 1. Αλλά και με αυτό ε, επιμένω ότι θα πρέπει σε περιφερειακό τουλάχιστον επίπεδο να είναι δυνατό να τηρηθεί το νήμιον 1 και γι' αυτό και τα βαλτικά κράτη θέλουν σε θέση να το τηρήσουν. Υπάρχει δυνατότητα αποθήκευση στη Λετωνία, Φερρυπίν, και ασφαλώ χρειάζεται καλύτερη διασύνδεση μεταξύ Δυτικής και Ανατολικής, ε, μεταξύ Ανατολής και Δύσης, αλλά υπάρχει δυνατότητα γι' αυτό, για την ε, αναστρεψιμότητα. Είναι ένα ζήτημα το οποίο πάντοτε με καταπλήσει στου όρου στου οποίου διεξάγεται η συζήτησή του, γιατί είναι πολύ μεγάλη πολυτέλεια για μα. Και μάλιστα κάποιο από του ε, πραγματογνώμονε, από του ειδικού, μου είχε ρωτήσει πώ είναι δυνατόν να συζητάτε τέτοιο ζήτημα. Πώ είναι δυνατόν να είναι και θέμα συζήτηση είναι τόσο ε, περιορισμένο το κόστος της εισαγωγής της αναστρεψιμότητας μέχρι 3 εκατομμύρια το πολύ για να γίνει η προσαρμογή ε, που δεν αξίζει τον κόπο και να τη συζητάμε. Ε, απλώς που, να πούμε ότι διαθέτουμε αυτά τα 3 εκατομμύρια και τελεία. Τίποτε άλλο δεν χρειάζεται ως συζήτηση. Δεν χρειάζεται να εξηγήσουμε γιατί το χρειαζόμαστε. Αυτά και σχέση με το 1 1 για τις εξουσίες Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Επιτροπή διεκδικεί βασικά δύο ειδών εξουσίες. Καταρχάς να ε, παληθεύει ότι είναι ε, κανονική η διαμόρφωση λειτουργία των εργοστασίων, των μονάδων παραγωγής ε, και Βεβαίω δεν θέλουμε να αποδυναμώσουμε τη δυνατότητα των κρατών μελών και τι επιχειρήσει, ε, οι οποίε προσπαθούν βέβαια σε ορισμένες χώρες προς κύριο τουρμέ να διατηρήσουν την κυριαρχή του θέση αλλά θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να είναι σε θέση να πει σε ένα κρατό κοιτάξτε αυτά που έχετε κάνει εδώ δεν είναι επαρκή, δεν μπορούν να ε, ασφαλίσουν, να διασφαλίσουν την κατάσταση ω προ την ενέργεια ανά πάσα στιγμή. Και θα πρέπει σε περίοδου κρίση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να είναι σε θέση να επαληθεύει ότι τα μέτρα που εισάγει ένα κρατό μέλο δεν στρεβλώνουν την εσωτερική αγορά όπω είδαμε το τον Ιανουάριο του 2009. Όλοι λοιπόν όσοι από εσά ανησυχούν ότι μπορεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να τυπώνει καινοτόμα ή νέα αιτήματα στα κράτη-μέλη, σα διαβεβαιώνω ότι δεν είναι αυτό. Απλώ θέλουμε να μην υπάρχει πρόβλημα ω προ τη ροή του φυσικού αερίου και την απρόσκοπτη λειτουργία τη εσωτερική αγορά και θα ήμουν ευγνώμων εάν ε, ε, υποστηρίζετε και εσεί αυτέ τι εξουσίε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όσον αφορά το όριο για την ε, κήρυξη του συναγερμού σε ευρωπαϊκό επίπεδο, εγώ προσωπικώ θα μπορούσα να δεχθώ και να μην υπάρχει ποσοτικό κατόφλι. Αρκεί να καθίσατε σαφέ ότι τη στιγμή που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα θεωρήσει ότι είναι κάτι ότι έχοντα αναλύσει και εξετάσει την κατάσταση εξωτικά θα είναι σε θέση να κηρύξει το συναγερμό. Από την άλλη όμως το 20% του ορίου που ορισμένα κάτι θεωρούν επαρκές είναι ασήμαντο πράγματι ασήμαντο ε, και πρέπει να υπενθυμίσω ότι στην προηγούμενη μεγάλη κρίση κύριε Ράνστοφ δεν είχαμε 20 ούτε 30% περικοπή των προμηθειών. 10% ήταν σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και προκάλεσε αυτή την κρίση. Για μένα λοιπόν πρέπει να είναι 10% το όριο, το κατόφλι καλύτερα, ή να μην αναγράφεται κανένα κατόφλι και να το κρίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επίσης θα θέλω να, να καταγράψω μια άλλη διάσταση, την εξωτερική διάσταση. Δεν ε, πιστεύω ότι υπάρχει πρόβλημα συνεργασίας μεταξύ του κυρίου Έτσιγκερ και της κυρίας Άστον. Δεν με ανησυχεί αυτή η διάσταση. Απλώς είναι σημαντικό να παραμείνει η απέτηση για τα κράτη-μέλη. Η απέτηση στα κράτη-μέλη να κοινοποιούν συμβάσεις με τρίτα μέρη μόλις ε, εγκαίρως. Αυτό είναι ε, όρος πραγματικής επικοινωνίας και έγκαιρης ενημέρωσης. Ε, βεβαίως μπορεί να μιλάτε για την ενημέρωση ex post, αλλά αυτό δεν σημαίνει ουσιαστική επικοινωνία. Θέλουμε πριν από τη σύναψη των συμβάσεων αυτών να κοινοποιούνται η συμβάσει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρόεδρε, αυτά και ελπίζω ότι με τι παρατηρήσει που απάντησα στι διάφορε ερωτήσει. Για τον κύριο Τούρμεν μόνο, η περιφερειακή συνεργασία δεν θα πρέπει να οδηγεί σε λιγότερο αυστηρή ρύθμιση, σε, πιο, σε χαλάρωση των ε, κανόνων και πάντως όχι σε παράβαση του όρου νήμιον 1. Και τέλος ο κύριος Βιδάλ να πάρει πάλι το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους που πήραν το λόγο για την ε, για τις προθέσεις τους, τις καλές τους προθέσεις να λύσουμε όλα τα προβλήματα που, είναι, που εκκρεμούν ακόμα. Οι συμβιβασμοί που θα προκύψουν πρέπει να είναι συμβιβασμοί που ανταποκρίνονται και στην πολυπλοκότητα των προβλημάτων. Δεν πρέπει να είναι συμβιβασμοί που να είναι συμβιβασμοί του να να ευχαριστήσουμε όλους χωρίς να ευχαριστούν με κανέναν. Πρέπει να είναι συμβιβασμοί που να ανταποκρίνονται σε πραγματικές αναγκαιότητες εξέβρεσης συμφωνίας και να πληρούν όρους που να απαντούν πλήρως στις ανάγκες μας. Παράδειγμα, η κυρία Μπαλεάν με την συνήθη της αποτελεσματικότητα και ευστοχία μας θύμισε ότι μπορεί να προκύψουν καταστάσεις όπου η κρίση του ανεφοδιασμού μπορεί να είναι μικρότερη του 10% του συνόλου της Ένωσης αλλά που για μία χώρα ή για μία ομάδα χωρών μπορεί να αποτελέσει καταστροφή και να χρειάζεται μια κοινοτική δράση για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε σε αυτό το πρόβλημα. Αντιθέτως, μια μεγάλη χώρα η οποία μπορεί να έχει μία, ένα πρόβλημα ανεφοδιασμού μεγαλύτερο του 10% μπορεί να έχει την ίδια δυνατότητα να βρει λύση από μόνο του και να μην χρειαστεί η κοινοτική έκτακτη ανάγκη για αυτή τη χώρα. Τώρα για την περιφερειακή εστίαση. Σίγουρα μπορεί να είναι δεσμευτική όταν υποκαθιστά ένα εθνικό σχέδιο αλλά μπορεί να είναι πολύ πιο θετικό όταν λειτουργεί συμπληρωματικά στα εθνικά σχέδια. Εμείς εδώ τώρα για τις εξουσίες της Κομισιόν δεν θέλουμε εμείς να δημιουργήσουμε ένα υπερ, υπερκράτος για την ασφάλεια του ανεφοδιασμού σε φυσικό αέριο. Αλλά η Κομισιόν πολύ ορθά λέει ότι πρέπει να έχει τη δυνατότητα για ορισμένα σημεία να προσανατολίζει την κοινοτική δράση, γιατί αλλιώς πραγματικά θα βρισκόμασταν στον αέρα. Εγώ πιστεύω λοιπόν ότι έχουμε πάρει καλό δρόμο και θα ήθελα να τονίσω για κάτι το οποίο συνειδητοποίησα μέσα από την ίδια την αρχή της συζήτησης για αυτόν τον κανονισμό. Εμείς πάντα λέμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να προσδίδει προστιθέμενη αξία στους πολίτες μας θα πρέπει να αποδεικνύει ότι για συγκεκριμένα πράγματα έχει τη δυνατότητα να βελτιώνει τους όρους ζωής και να απαντάει στα προβλήματα των Ευρωπαίων πολιτών. Αυτός ο κανονισμός αποτελεί παραδειγματικό, πα, ε, απτό παράδειγμα για την πραγματικότητα αυτής της ε, άποψης. Έχει λοιπόν νόημα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας ευχαριστώ και έτσι κλείνουμε το σημείο αυτό στην ημερήσια διάταξη και με, με κάποια καθυστέρηση να περάσουμε στις ε, ψηφοφορίες. Έχουμε αρκετές ψηφοφορίες σήμερα. Να προσπαθήσουμε να δούμε αν λειτουργεί το τεχνικό τμήμα της υπόθεσης καταρχάς. Δεν ξέρω τι πρόβλημα υπάρχει. Δεν ξέρω αν υπάρχει πρόβλημα. Έχετε όλοι μαζί τις κάρτες σας. Να κάνουμε μία δοκιμή. What happens? correct? Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Συνάδελφοι, λίγη ησυχία παρακαλώ για να ακούμε ένα τον άλλον και για να ξεκινήσουμε τις ψηφοφορίες. Όσοι θέλουν να συζητήσουν, παρακαλώ έξω. Όσοι θέλουν να ψηφίσουν, να κάτσουν μέσα στην αίθουσα. Ύστερα, να κάνουμε μια δοκιμαστική ψηφοφορία, να δούμε αν λειτουργούν τα μηχανήματα. Παρακαλώ ψηφίστε για το αν θα πρέπει στο μέλλον να ξεκινάμε στην ώρα μας τις συνεδριάσεις. Ναι, όχι οι αποχές. Ε, μα δεν έχω τίποτα άλλο να πω για να ψηφίσουμε. Σας παρακαλώ ψηφίστε. Πέρας ψηφοφορίας. Ωραία, σας ευχαριστώ. Λειτουργούμε. Εντάξει, εντάξει. Okay. Το ξεχάσατε, ξεχάσατε την κάρτα σας. Τι κάνετε. Την άλλη φορά να έρθετε λίγο πιο νωρί. Αυτό λοιπόν, εντάξει. Ε, δύο μηχανήματα έχουν πρόβλημα. Παρακαλώ τον τεχνικό να κοιτάξει τα δύο αυτά μηχανήματα στην δεύτερη σειρά. Μία παρατήρηση επί της διαδικασίας από τον κύριο Ντί. Merci, Monsieur le Président. Pour des motifs d'urgence. Πρόεδρε, για λόγου Ενημερωθήκαμε ότι είμαστε υποχρεωμένοι να καταθέσουμε τι τροπολογίε στα αγγλικά, επειδή δεν υπήρχε χρόνο. Διαμαρτύρομαι επισήμω. Τροπολογία είναι κοινοβουλευτικό δικαίωμα είμαστε εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Υποτίθεται ότι εκπροσωπούμε κράτη τα οποία ε, σε παγκόσμιο επίπεδο πρωτοπορούν ε, νομοθετώντας μέσω των ερετών τους εκπροσώπων και σε όρους δημοκρατίας και πρέπει να έχουμε το δικαίωμα ο καθένας να μιλάει και να γράφει στην αμυντρική του γλώσσα. Κύριος Λάγκη. Θέλω και εγώ ρητά να υποστηρίξω τον συνάδελφο και τις θέσεις του. Και ύστερα να σας ανακοινώσω ότι και εγώ το υποστηρίζω αυτό αφενός. Αφετέρου όμως, κάναμε μια συμφωνία εδώ στην Επιτροπή μας και αυτό ε, θα πρέπει να το τιμήσουμε τη συμφωνία που κάναμε πριν από κάποιες συνεδριάσεις για αυτό το θέμα της ημερήσιας διάταξης, για το θέμα αυτό που το συζητούσαμε. Δεν ξέρω αν ήταν όλοι παρόντες, αλλά συμφωνήσαμε και συζητήσαμε επειδή ήταν εξαιρετικές δυσκολίες ε, για να ολοκληρώσουμε τη διαδικασία εγκαίρως, είχαμε παρακαλέσει την Επιτροπή Πολιτισμού να αναβάλει την ε, όλη διαδικασία προκειμένου να τα καταφέρουμε, αλλά δεν υπήρχε άλλη δυνατότητα και γι' αυτό συμφωνήσαμε και συμφώνησαν όλα τα μέλη της Επιτροπής που ήταν παρόντα στη συνεδρίαση αυτή. Ε, λυπάμαι, τι να κάνω. Επί της αρχής, 100% δίκιο σας δίνω. Αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση ήταν μια συμφωνία την οποία πρέπει να τιμήσω πλέον και να τηρήσω. Ε, δεν μπορούμε να αλλάζουμε κάθε εβδομάδα αυτού του κανόνε, να γίνει. Έτσι αποφασίσαμε από κοινού, αυτό και θα κάνουμε. Ίσως όμω να μπορέσουμε να βρούμε μια λύση για τη συγκεκριμένη περίπτωση που έχετε πρόβλημα. Ο κύριος Οντί. Εγώ θα ήθελα να ξέρω, Πρόεδρε, ποια είναι η νομική βάση μια τέτοια συμφωνία. ένα σοσιαλιστής Γάλλος ε, βουλευτή είπε νομικά έχετε άδικο γιατί πολιτικά είστε με μειοψηφία. Δεν κατάλαβα εγώ από πού και ως πού ένας βουλευτής να μην μπορεί να καταθέτει τροπολογία στη γλώσσα του. Η γραμματεία μπορεί να απαντήσει παρακαλώ. Euh, Μα υπάρχουν ειδικέ παρεκκλήσει που εφαρμόζονται καταρχήν στην, ε, βασικά μάλλον στην Ολομέλεια. Για κανονισμούς που δεν ε, κατετίθενται σε όλες τις γλώσσες και υπάρχουν ε, επίσης ε, και όροι που επιτρέπουν ε, στους βουλευτές να προβάλλουν αντιρρήσεις ε, στην απόφαση του Προέδρου. Αλλά ο κανονισμός δεν λέει τίποτα για αυτού του είδους τις διατάξεις. Ωραία λοιπόν. Να ακολουθήσουμε τη διαδικασία που είχε αποφασίσει η Επιτροπή μας τότε θα προσπαθήσουμε να βρούμε μια λύση ωστόσο για το συγκεκριμένο αυτό πρόβλημα. Μιλάμε τώρα λοιπόν για την έκθεση Beauty Coffer καταρχάς. Έχετε μπροστά σας τα απαραίτητα έγγραφα. Νομίζω ότι... Α, συγγνώμη, να ψηφίσουμε την τροπολογία 1. Ίσως να ψηφίζουμε διανάταση ισχυρό και αν υπάρχουν αμφιβολίες να ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Τροπολογία 1. Υπέρ κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 2, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται η 3 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα, υπέρ, α, συγγνώμη, καταπληκτή. Να το ελέγξουμε για το πρώτο τμήμα, μάλιστα. Οκ, να ε, ψηφίσουμε ηλεκτρονικά το πρώτο τμήμα. Ηλεκτρονικά, παρακαλώ. Έναρξη ψηφοφορία. Α, έχουμε έναν από το ΕΛΚ. Δύο από το ΕΛΚ που δεν πρέπει να ψηφίσουν. Δύο ψήφους παραπάνω από το ΕΛΚ. Noch einer. E Ένας ακόμα περισσεύει. Τώρα μάλιστα, εντάξει. Πέρας. Αποτέλεσμα 13. Α, ναι, υπέρ, 38 κατά. Απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα. Α, είπαμε ότι καταπίπτει. Και περνάμε στην τροπολογία 5 και αυτή σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Με προφορική τροπολογία, παρακαλώ. Υπέρ. Κατά λοιπόν τώρα. δεν είναι σαφές. Έλεγχος παρακαλώ ηλεκτρονικά. Ε, Για την προφορική τροπολογία. Μόνο την προφορική τροπολογία. Ηλεκτρονικά παρακαλώ. Abstimmung eröffnet. Abstimmung geschlossen. Πέρας ψηφοφορίας παρακαλώ. Εγκρίνεται. Ο κύριος Οντί. Διαδικαστικό. Συγγνώμη κύριε Πρόεδρε, αλλά πιστεύω ότι δεν ψηφίσαμε την 4. Σας ευχαριστώ. Δικό μου λάθος. Να ψηφίσουμε μόνο το δεύτερο τμήμα πρώτα και μετά να περάσουμε στην τροπολογία. Στο δεύτερο τμήμα τις πέντε παρακαλώ. Α, όχι, λέει ο Πετρος. Alles weg, alles Okay. Καταπίπτει. Ωραία λοιπόν. Να περάσουμε στην τροπολογία 4. Και συγγνώμη, δικό μου σφάλμα λέει ο πρόεδρος. Να ψηφίσουμε την τροπολογία που έχουμε μόνο στα γαλλικά. Αν μου επιτρέπετε να την ε, διεκπαιρεώσουμε τροπολογία για να τη μεταφράσουμε. Εντάξει. Υπάρχουν αντιρρήσεις. Ε, Κύριε Πιτεκόφερ, σας παρακαλώ, ξανασκεφτείτε το, λέει ο Πρόεδρος. Μα Πρόεδρε, η τροπολογία αυτή δεν μου έχει δοθεί στα αγγλικά ως εισηγητή και είχαμε συζητήσει όλα να υποβληθούν στα αγγλικά. Ε, μα δεν ξέρω αρκετά γαλλικά για να καταλάβω τροπολογία ολόκληρη στα γαλλικά. Είχε ο συνάδελφος που υπέβαλε την τροπολογία να έρθει σε επαφή μαζί μου και να μου την εξηγήσει, να μου την εξηγήσει. δεν το έκανε, ε, άρα δεν βλέπω γιατί να ψηφίσουμε τώρα κάτι το οποίο έτσι παρουσιάζει ad hoc ο συνάδελφος. Δεν μπορεί να υπάρχει ε, πραγματικά να σχηματίσουμε μια ολοκληρωμένη άποψη με τον τρόπο αυτό. Ο Πρόεδρος, η πρότασή μου είναι να την υποβάλουμε ως προφορική τροπολογία. Στην περίπτωση αυτή θα μεταφραστεί. Αλλά αν υπάρχουν αντιρρήσεις, ε, ο κανονισμός είναι σαφής. Εγώ απλά πρότεινα μία μικρή απόκληση <coughs> από τον κανονισμό. Ο κύριος Λάνη ζητάει το λόγο. Αν συμφωνήσουμε, εφόσον συμφωνήσαμε στα αγγλικά και δεν επιτρέπουμε την παράλληλη, την ταυτόχρονη διερμηνία, προτείνω να διακόψουμε την ψηφοφορία και να φροντίσουμε την επόμενη φορά να υπάρχουν όλες οι γλωσσικές ε, εκδόσεις ε, των τροπολογιών. Κύριε Σοντή. Κύριε Πρόεδρε, ήθελα να συναντήσω εγώ τον ε, εισηγητή, είχαμε όμως πολλές συναντήσεις με τη γαλλική αντιπροσωπεία και δεν κατάφερα να τον δω. Λοιπόν, πρόταση. Αν οι συνάδελφοι δεχθούν αυτή την τροπολογία, θα σας το διαβάσω, θα ακούσετε τη διερμηνία και μετά θα αποφασίσετε. Κυρία Κόμι, Εγώ δεν συμφωνώ. Νου. Ο συνάδελφος um, with... Ευχαριστώ, Πρόεδρο. Πρόεδρε. Αν ακολουθήσουμε την παράδοση της Επιτροπής, θα πρέπει να ε, κοιτάξουμε την ε, τροπολογία ως προφορική τροπολογία για να μας τη μεταφράσουν ε, οι διερμηνείς. Και έτσι θα ακούσουν όλοι οι συνάδελφοι στη μητρική τους γλώσσα. Α ακολουθήσουμε λοιπόν αυτή την παράδοση, προτείνω εγώ. Κύριε Μπιτικόφερ, εξ όσων γνωρίζω, ο κανονισμός προβλέπει ότι κάθε μέλος τη Επιτροπής μπορεί να υποβάλει ένσταση για τέτοια θέματα. μπορεί, ε, είμαι δεθυμένος <coughs> να κάνω μια υποχώρηση εφόσον ζήτησε συγγνώμη ο υποβάλλον της τροπολογίας, μάλιστα. Ωραία. Κύριε Οντί, θα διαβάσετε παρακαλώ την ε, τροπολογία σας στα γαλλικά. Με αργό ρυθμό παρακαλώ για να την ακούσουμε καλά και από τις καμπίνες. Για να ακούσουμε λοιπόν την τροπολογία και να την ψηφίσουμε. Σας ευχαριστώ που δείξατε πνεύμα συμβιβασμού και καταφέραμε να συμφωνήσουμε. Κύριε Οντί. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε να ευχαριστήσω πρώτα από όλα τον συνάδελφο. Λοιπόν, καλεί την Κομισιόν να εγκρίνει μια ολιστική και συνολική άποψη ούτω ώστε να έλξει την Ευρώπη για την ανάπτυξη, την απασχόληση και καλεί την Κομισιόν να ξεκινήσει με το Κοινοβούλιο μία συζήτηση για την αποτελεσματικότητα της πολιτικής του ανταγωνισμού και να διασφαλίσει ότι η τωρινή πολιτική αντιτράστε η οποία βασίζεται σε ψηλά πρόστιμα που υπολογίζονται στο τζίρο των επιχειρήσεων χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα πραγματικά αποτελέσματα είναι ρήψο κίνδυνα και μπορούν να οδηγήσουν στην εξαφάνιση των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων εις βάρος της απασχόλησης. Και αναρωτιέται αν η εφαρμογή των προστήμων δεν θα πρέπει να αποσυνδεθεί από την προσωπική στάση και συμπεριφορά των επιχειρηματιών από την ίδια την επιχείρηση. Όλα αυτά τα διάβασε με τρομερή ταχύτητα ο μιλητής, ο διερμηνέα δεν κατάφερε να δώσει λέξη προς λέξη την τροπολογία όπως ένας μεταφραστής θα έκανε. Πολύ για τη μετάφραση λέει ο Πρόεδρος. Μπορούμε λοιπόν να ψηφίσουμε υπέρ της τροπολογίας περιθμών 4. Κατά. Απορρίπτεται. Και σας ευχαριστώ. Η υπαριθμόν 6 υπέρ παρακαλώ. Κατά της υπαριθμόν 6. Αποχές. Απορρίπτεται. 7. Σε τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. Οχτώ. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ε, δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 9 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 10 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 11 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 12 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 13 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 16 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 15 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται 14 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται Επτά, Πρώτο τμήμα της επτά, Υπέρ. Όχι, στην παράγραφο επτά, Αρχικό κείμενο. Πρώτο κομμάτι υπέρ. Κατά. Αποχές. Να επαληθεύσουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. πέρα τη ψηφοφορία. Εγκρίνεται. 17 υπέρ. Όχι, καταπίπτει. Καλώς 18 τότε. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Το σύνολο της προτάσεως παρακαλώ υπέρ. καλός ηλεκτρονικός ε, ηλεκτρονική ψηφοφορία, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα της ψηφοφορίας. Ένας από το ΕΛΚ περισσεύει. Πέρα της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται λοιπόν στην προσεχή ψηφοφορία τώρα και συγχαρητήρια. Έκθεση Βαλιάν. λίγο πιο περιπλοκή. Πολλές προφορικές τροπολογίες παρακαλώ να μας βοηθήσετε. 27 28 και προφορική τροπολογία. 27-28 προφορική τροπολογία. Ποιος είναι υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές εγκρίνεται και πάμε στη συμβαστική υπαριθμών 1 υπέρ κατά αποχές. Κύριε Πρόεδρε, είχα ζητήσει το λόγο πριν να ξεκινήσει η ψηφοφορία, αλλά δεν με είχατε δει. Ναι, κύριε Τιτσό. Ήθελα να σημειώσω ότι στην υπαριθμόν 50 ε, υπαριθμών 50 δεν καλύπτεται από την προφορική τροπολογία υπαριθμών 1. Η 50 δεν περιλαμβάνεται στο κείμενο του συμβασμού. Παρακαλώ να το σημειώσετε. Ναι, αλλά φαίνεται ότι έχουν κάνει Συμβαστική πρόταση. Το έχουν χειριστεί ως συμβασμό οι συντονιστές από τις ομάδες. Γι' αυτό άμα δεν σας ε, βολεύει μιλήστε με τον εκπρόσωπο της ομάδας σας. Τίποτα άλλο δεν μπορούμε να κάνουμε προς το παρόν. Κυρία Βαλιάν. Δεν καλύπτεται από τη συμβαστική η 50, αλλά εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογή της. Κατά με είναι απλό, πολύ απλό. Also, ähm, das sind manchmal... Ναι, μερικές φορές το έχουμε το πρόβλημα αυτό κυρία Τιτσάου, το έχω δει και εγώ στο παρελθόν. Πρέπει να κοιτάμε πολύ προσεκτικά την, ε, το περιεχόμενο. Ίσως έχουμε τη δυνατότητα στην συνολομέλεια να το ξαναδούμε. Η ένα λοιπόν εντάξει, η δύο συμβαστική υπέρ, κατά Αποχές. Με πλειοψηφία λοιπόν. 54 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 55. Προφορική τροπολογία. Ο μπλοκ μαζί με τη συμβαστική 4. Πολύ περίπλοκα είναι. 55 και συμβαστική 4. Μαζί. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κατά. Αποχές. Εγκρίνεται 56. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 57 υπέρ. Μέσα με την Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική υπαριθμών 3 με προφορική τροπολογία για την 82 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται οι άλλες καταπίπτουν πάμε στην 11 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 66 υπέρ 65, όχι λυπούμε, 63, ζητώ συγγνώμη, είναι πολλές του κυρίου Γκίρεκ, 63 του κυρίου Γκίρεκ ψηφίζουμε τώρα, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται, 65 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται, 66 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται, συμβαστική, 3 υπέρ αποχές εγκρίνεται 96 υπέρ 69 ε, συγγνώμη υπέρ Άρχεται η ψηφοφορία κατά εγκρίνεται στην 70 έχουμε μια προφορική παρατήρηση που έχει καλύψει το πρόβλημα. 71, 71 υπέρ, κατά. Αποχές, ε, απορρίπτεται. 72, πρώτο κομμάτι. Ευχαριστώ, κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 73 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 74 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 75 και 76 ταυτόσιμες υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 77 και 78 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 12 υπέρ κατά Αποχές εγκρίνεται. 79 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 80. Δεύτερο τμήμα με προφορική τροπολογία. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 13 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 81 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Ε, παριθμόν 2 της Επιτροπής Περιβάλλοντος υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Η 14 και η MV3 υπέρ Κατά. Ευχαριστώ. Αποχές. ε, NV4 υπέρ. Κατά. Αποχές. Έρβη NV5 υπέρ. Κατά. Ας επαληθεύσουμε. Οι πέντε της NV ε, ελέγχουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 55 υπέρ. Κατά. 85 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 86 ε, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 15 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 87 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτωτα. 16 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται 88 και 90 μαζί υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 89 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 5 υπέρ με en μάλλον μαζί με την προφορική τροπολογία για την 91 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται NV6 υπέρ κατά αποχές απόρριπτεται 19 υπέρ κατά Αποχές εγκρίνεται 95 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται 20 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται 96 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 6 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 99 με προφορική τροπολογία υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 101 τώρα προφορική τροπολογία, με προφορική τροπολογία υπέρ. Κατά. Ας επαληθεύσουμε παρακαλώ. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 7. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η 105 με προφορική τροπολογία υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 22 υπέρ. Κατά Αποχές εγκρίνεται. 108 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 109 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 110 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 112 υπέρ. Κατά. Αποχές Ας επαληθεύσουμε. 112. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία πάλι. Δεν δουλεύει. Ναι, να το ξανακάνουμε, εντάξει. Υπέρ, κατά, τι θέλετε. 29, 34 εγκρίνεται. Τώρα πάμε στην 112, 113 μάλλον υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 114 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 115 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 116 υπέρ κατά αποχές 100, ε, εγκρίνεται 117 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 118 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 25 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 119 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 120 υπέρ κατά αποχές Απορρίπτεται 121 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται 122 προφορική τροπολογία. Με προφορική τροπολογία. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 123 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 26 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 126 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 127 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 128 υπέρ κατά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 Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 7 της ένβη υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 132 έχει αποσυρθεί 136 ε, υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 134 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 135 υπέρ Κατά. Αποχές απορρίπτεται 29 ε, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται 30 καταπίπτει. Και τώρα έχουμε την υπαριθμόν 1. 1 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται στην 31 προφορική τροπολογία υπέρ κατά αποχές ας το επαληθεύσουμε παρακαλώ την 31 άρχεται η ψηφοφορία πέρας καταπίπτει υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ευχαριστώ 33 υπέρ καταπίπτει καλά 34 υπέρ κατά Αποχές. Ας επαληθεύσουμε. Ναι, ε, ε, ψηφίζουμε την 34 παρακαλώ. Πέρα στις ψηφοφορίας εγκρίνεται. Η 34, πάμε σε 35, σε τμήματα. Πρώτο, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά να επαληθεύσουμε παρακαλώ το δεύτερο τμήμα της 35 άρχεται η ψηφοφορία πέρας αποτέλεσμα εγκρίνεται τρίτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 36 υπέρ κατά Αποχές εγκρίνεται. Η πρώτη τη Επιτροπή Περιβάλλοντο, Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Σε τμήματα η 37. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα έχει αποσυρθεί. Υπάρχει μόνο δύο. Παρακαλώ υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται 39 πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα έχει αποσυρθεί συμβαστική 10 ε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται περνάμε στην 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 42 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 43 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 7 υπέρ κατά 8 ε, εγκρίνεται 44 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ο κύριος Τσούρμες έχει το λόγο Ψηφίζουμε την αιτιολογική. Ψηφίσαμε την προφορική επί ε, της αιτιολογικής σκέψης 48. Α, ναι, με συμβιβαστική. Μάλιστα, μάλιστα. Ευχαριστώ. Είσαστε εντάξει, κύριε Πρόεδρος. Σα... 45 κατά αποχές εγκρίνεται 46 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται είχε κατά 47 και τώρα μπορούμε να ψηφίσουμε το σύνολο ηλεκτρονικά παρακαλώ άρχεται η ψηφοφορία πέρας της ψηφοφορίας εγκρίνεται και συγχαρητήρια και τώρα πάμε στη ψηφορία για το νομοθετικό ψήφισμα. Ηλεκτρονικά ή όχι. Ηλεκτρονικά και πάλι ψηφοφορία για το νομοθετικό ψήφισμα, αρχή ψηφοφορία, πέρας ψηφοφορίας, αποτέλεσμα, όχι έκλεισε. Ναι, το ίδιο αποτέλεσμα, ευχαριστώ πολύ. Και περνάμε τώρα στο Ευρωπαϊκό, στο επόμενο θέμα του συναδέλφου Ένσιου. Και αυτή, και αυτή η ψηφοφορία θα είναι λίγο περίεργη. Τροπολογία 2, υπέρ. Κατά. Για τη 2 παρακαλώ, ποιος είναι υπέρ. Μια φορά ακόμη. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. 3. Κατά. Αποχές Εγκρίνεται. Στην 4 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Να, και τις αποχές ξέχασα. 5 υπέρ. Με την προφορική τροπολογία. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Στο 6 δεύτερο τμήμα παρακαλώ. Για το 6, δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Και αυτό λοιπόν εγκρίνεται. 7. Με την προφορική τροπολογία του κυρίου Τσουκαλά. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 8. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η 9. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η 10. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η 11. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 12. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η 13. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η 14 με την προφορική τροπολογία. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. Αποσύρεται η 15 στην 16. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. Η 17 με προφορική τροπολογία. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. 18. Υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. 19 σε δύο τμήματα, πρώτο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Το δεύτερο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 20 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 21 υπέρ, κατά, Αποχές εγκρίνεται. 22 με προφορική τροπολογία. Υπέρ. Κατά. άποχέ. εγκρίνεται. 23 υπέρ. Κατά. Αποχέ. εγκρίνεται. 24 υπέρ. Κατά. Αποχέ. εγκρίνεται. 25 υπέρ. Κατά. Αποχέ. εγκρίνεται. 26 υπέρ. Κατά Άποχες. Εγκρίνεται. 27 υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. Η 1 υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. Äh, Έχουμε ένα, μια αίτηση των πρασίνων, το πρώτο τμήμα Τη τροπολογία 6 να ψηφιστεί. Ενώ οι συνάδελφοι είχαν ε, συμφωνήσει να μην ψηφιστεί, να αποσυρθεί αν ε, εγκριθούν οι 4 και οι 5, αλλά εφόσον επιμένουν να την ψηφίσουμε και αυτήν λοιπόν. Απλά να συμφωνήσουν οι ομάδες τι θα κάνουμε, γιατί δεν έχει προβλεφθεί κάτι τέτοιο. Θα ψηφίσουμε τώρα το πρώτο τμήμα της 6. Αντίθετα μετά όσα λέει ο κατάλληλος ψηφοφορίας. Υπέρ. Κατά. Άλλη μία φορά παρακαλώ. Ηλεκτρονικά. Το πρώτο τμήμα της 6. Ηλεκτρονικά παρακαλώ. Πρόβλημα. Ναι, θα μπορούσατε να μας εξηγήσετε και πάλι τι ακριβώς ψηφίζουμε. Ναι, να τα εξηγήσω άλλη μια φορά, λέει ο Πρόεδρος. Από την τροπολογία 6, το πρώτο τμήμα. Είχαν συμφωνήσει μεταξύ τους οι ομάδες να το θεωρήσουν διακπεραιωμένο από αυτή που λέει to improve the management. Θεωρούταν λοιπόν, είχε θεωρηθεί ότι θα κατέπιπτε εφόσον είχε εγκριθεί 4 και 5. Ωστόσο οι πράσινοι ζητούν τώρα να ψηφιστεί παρόλα αυτά. Καταλάβατε λοιπόν τι έγινε. Το improve the management. Να το προσθέσουμε ή όχι. Ηλεκτρονική ψηφοφορία παρακαλώ. Έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας. Εγκρίνεται. Και τώρα περνάμε στην τελική ψηφοφορία. ηλεκτρονικά παρακαλώ. Έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας. Το αποτέλεσμα το βλέπετε. Συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια. Επόμενη ψηφοφορία. για την εγκατάσταση του τηλεσκοπίου ELT. Εγκρίνεται. Δεν ξέρω, υπάρχουν ε, ψήφοι κατά. Όχι, φυσικά, όλοι είναι υπέρ. Μα φανταστικά τα πήγε ο εισηγητή σε αυτήν την έκθεση. Και περνάμε στο επόμενο θέμα, η ψηφοφορία Τσερσνόφσκι, την οποία την βάλαμε στην ημερήσια διάταξη. Θα ψηφίσουμε λοιπόν Τροπολογία 1. Συμβαστική τροπολογία 1. Υπέρ. Ευχαριστώ κατά. Άποχες. Αποφασίστηκε. Λοιπόν, υπέρ. Συμβαστική 2. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. Η 27. Υπέρ. Κατά. Άποχες εγκρίνεται. Συμβαστική τρία υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Καταπίπτει. Στην 28 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η 9 υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. 11 υπέρ. Κατά. Άλλη μια φορά παρακαλώ για την 11 υπέρ. Για την 11 παρακαλώ υπέρ. Για την 11 υπέρ παρακαλώ για την 11 κατά αποχές εγκρίνεται 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Η 29 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 15 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 1 υπέρ. Κατά. Αποχέ εγκρίνεται. Η 2 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. και η τρία εντάξει. Στην πέντε λοιπόν, στην βασική πέντε. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Πέντε, υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. Έξι, υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. Και τώρα περνάμε στην ε, τελική ψηφοφορία για το σύνολο του κειμένου, παρακαλώ. Α, όχι, συγγνώμη, το κείμενο όπως τροποποιήθηκε. Ηλεκτρονικά, όχι, το χρειάζεται. Ωραία. Υπέρ, παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Με μεγάλη πλειοψηφία εγκρίνονται λοιπόν και περνάμε τώρα στο... Δεν θα ψηφίσουμε το νομοθετικό, την νομοθετική πρόταση γιατί ακόμα συζητιέται. Ολοκληρώσαμε λοιπόν και το θέμα αυτό και έτσι κλείσαμε τις ψηφοφορίες, κυρίες και κύριοι. Ε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, αλλά παρακαλώ να μείνετε στην αίθουσα γιατί έχουμε και άλλα θέματα και περνάμε στο 9. Την κατάρτιση μιας νέας ευρωπαϊκής ατζέντας για την ψηφιακή τεχνολογία για την Ευρώπη. Έχουμε τα έγγραφά μας. Θα γίνει μια πρώτη συζήτηση σήμερα. Η κυρία Ντελκαστήγιο είναι η συγκήτρια και θα της δώσω το λόγο πάρα αυτά. Αλλά σας παρακαλώ κυρίες και κύριοι, μα συνάδελφοι, σε περίπτωση που έχετε επίγουσε συζητήσει. περάστε παρακαλώ έξω. Έχει πολύ χώρο. Ύστερα. Μα σας παρακαλώ, λίγο ησυχία. Σας ευχαριστώ πολύ. Και τώρα θα δώσω το λόγο στην κυρία Ντέλ Καστίγιο. Και θα ήθελα επίσης να καλωσορίσω τον κύριο Κολασάντη ως εκπρόσωπο των ομάδων. Ε, να περιμένουμε μισό λεπτό γιατί είναι δύσκολο και έχει πολύ φασαρία. Why is it so complicated to go out? γιατί είναι τόσο περίπλοκο να βγει ο κόσμο έξω. Σας παρακαλώ, γρήγορα τουλάχιστον. Somebody announced me. Äh, ε, Κυρίε και κύριοι, έχουν ζητήσει το λόγο συνάδελφοι. Καταρχάς, να δώσουμε το λόγο στην κυρία Δελκαστήγιο. Έχετε το λόγο, να μα ενημερώσετε. Ε, Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Λοιπόν, ε, στο τέλος της, σημερινή, της ε, συνεδρίασης της Πέμπτης θα πρέπει να μιλήσουμε για την ε, ψηφιακή ατζέντα που επεξεργάστηκε το Κοινοβούλιο κατόπιν αιτήματος της Κομισιόν με μένα φυσικά η συγκήτρια και έχοντας ως στόχο πριν δηλαδή η Κομισιόν μας παρουσιάσει το έγγραφό της για την ψηφιακή ατζέντα για την Ευρώπη, το Κοινοβούλιο να έχει εκφράσει τη δική του και τα κράτη-μέλη και το Συμβούλιο να μπορέσουν να λάβουν υπόψη τη θέση του Κοινοβουλίου όταν φυσικά καταλήξουμε στην οριστική μας ε, ε, άποψη. Δεν θέλω εγώ να επεκταθώ ε, λέγοντας πόσο αποφασιστικές και σημαντικές είναι οι τεχνολογίες ε, επικοινωνίας και πληροφόρηση σήμερα που ρυθμίζουν ε, συνολικά την κοινωνική και οικονομική ζωή. Σήμερα βρισκόμαστε στην αρχή μίας ψηφιακής ε, ιστορικής περίοδου. Τι πρέπει να επιλέξουμε, το business as usual ως μέθοδο ή θα πρέπει εμείς ε, να επιταχύνουμε αυτό το βήμα προς την ψηφιακή εποχή. Έχουμε εμείς ε, παραδείγματα σε άλλες ε, φάσεις της πληροφορικής επανάστασης. Εμείς ε, περνάμε από την εποχή του ατόμου στην εποχή του byte. Χρειάζεται λοιπόν να έχουμε υπόψη σε αυτό το πέρασμα εποχής, σε αυτή την αλλαγή ιστορικής φάσης, το, τον άνθρωπο, και την ατομικότητα του κάθε ανθρώπου. Η Κομισιόν, τα κράτη-μέλη, ε, όλοι συζητούν για μια ψηφιακή ατζέντα για το πώς μπορούν να κάνουν ένα βήμα παραπάνω λαμβάνοντας ε, μέτρα δράσης ε, και παρακολούθησης ούτως ώστε η Ευρώπη να μπορέσει να επωφεληθεί απόλυτα από αυτήν την ψηφιακή επανάσταση. Αν θα έπρεπε να ορίσω τι είναι μία ψηφιακή ατζέντα είναι ένα σύνολο προσανατολισμών που θέλουν να προσεγγίσουν ορισμένους στόχους μέσα από ειδικέ δράσεις και μεθόδους παρακολούθησης αυτών των δράσεων ούτω ώστε να υποφεληθούμε το μάξιμουμ από την ψηφιακή επανάσταση. Διότι ή θα τα εκμεταλλευτούμε όλα αυτά τα πλεονεκτήματα ή αλλιώς θα μείνουμε πίσω απέναντι σε άλλες γεωπολιτικές ζώνες ε, του πλανήτη ε, που θα πάρουν την πρωτοκαθεδρία. Αυτό το οποίο παρουσιάζω εγώ σήμερα λοιπόν είναι αυτή η ατζέντα 2015 παπάκι ΕΟΥ το 2005, 2015 ε, για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο πυρήνας αυτού του σπιράλ που σας δίνω εδώ ως γραφικό σχήμα είναι ο άνθρωπος που θα πρέπει να έχει τις ειδικέ ικανότητες, δυνατότητες πρόσβασης από οπουδήποτε, ταχύτητα πρόσβασης και επίσης δικαιώματα που θα τους προστατεύουν και στη δυνατότητα πρόσβασης αλλά και στην ασφάλεια ούτως ώστε να μπορούν να λειτουργήσουν σε αυτό το νέο ψηφιακό σενάριο. Μέσα λοιπόν από αυτόν τον κεντρικό πυρήνα αναπτύσσονται άλλες πλευρές που είναι απόλυτα ουσιαστικές για να μπορέσουμε να προωθήσουμε αυτή την ψηφιακή κοινωνία στην Ευρώπη. Καταρχήν, τι θέλουμε να προσεγγίσουμε. Είναι η ενιαία ψηφιακή αγορά, ενιαία και ανοιχτή, όπου η ανταγωνιστικότητα παίζει ουσιαστικό ρόλο, διότι η αγορά η ανταγωνιστική θα είναι η Αλλιώς δεν θα πετύχει στο στόχο της ε, ε, για την παροχή ε, αγαθών και υπηρεσιών προς τους πολίτες, διότι δεν θα υπάρχει ελευθερία επιλογής και αυτό φυσικά προδικάζει την αγορά και την οικονομία. διότι περιορίζονται οι δυνατότητες ανταγωνισμού παγκοσμίως. και πρόκειται για ένα χώρο με 500 εκατομμύρια ενδυνάμει καταναλωτές. Και υπάρχει και ένας τελευταίος κύκλος αυτό το σπιράλ που μας οδηγεί στην κοινωνία. Δηλαδή, ευημερία, στόχος. Λοιπόν, η ευημερία. Για να την πετύχουμε χρειάζεται αριστείο, αριστεία στην έρευνα και παροχή ανταγωνιστικών δυνατοτήτων στη βιομηχανία μας και κυρίως στις ΜΜΕ που αποτελούν και τη βάση του βιομηχανικού ιστού και που παίζουν σημαντικότατο ρόλο στην πρόθεση της ψηφιακής κοινωνίας. Πρέπει λοιπόν οι ΜΜΕ να καρποθούν όλα αυτά τα ωφελήματα γιατί αλλιώς δεν θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Αυτά λοιπόν στο γραφικό σχήμα. Και έχω και άλλα στοιχεία τα οποία θεωρώ ότι είναι απαράβατα για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στην ψηφιακή πρόοδο αφενός πολιτική leadership δηλαδή Η ψηφιακή ατζέντα θα πρέπει να είναι η διοκτησία της πολιτικής ευρωπαϊκής έκφρασης από την τοπική αυτοδίκηση ως την ανώτατη αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή η πολιτική οργάνωση της Ένωσης να είναι ιδιοκτήτρια αυτών των στοιχείων, γιατί αλλιώς δεν θα μπορέσουν να αναπτυχθούν. Χρειάζεται επίσης ορατότητα πρέπει να ληφθούν ας πούμε αποφάσεις ούτω ώστε να γίνεται ενημέρωση, να έχουμε ας πούμε μία εβδομάδα κάθε χρόνο αφιερωμένη στην ψηφιακή ατζέντα. και ενημέρωση για τους στόχους του καθενός σχετικά με την ψηφιακή ατζέντα. Ας πούμε, η κάθε προεδρία να παρουσιάζει ποιο είναι το σχέδιό της. Ας πούμε, καταρχήν η Ισπανική Προεδρία και μετά όλες οι υπόλοιπες. Πρόκειται για στοιχεία κλειδί. Πού? Ξεκινάνε πρώτα από τον άνθρωπο διότι σε αυτή τη φάση επανάστασης πρέπει να ενδυναμώσουμε τα άτομα όχι μόνο ως προς την απόκτηση της γνώσης αλλά και ως προς τον τρόπο εφαρμογής αυτής της γνώσης δηλαδή ικανότητα χρήσης, ε, παροχή δικτύων Όλοι δηλαδή να μπορούν να εκμεταλλευτούν απόλυτα όλες τις ευκαιρίες αυτής της ε, ψηφιακής επανάστασης. που βρίσκεται στα σπάργανα υπό κάποια έννοια. Θα μπορούσαμε εν μέρη να συγκρίνουμε την ψηφιακή επανάσταση με τη βιομηχανική επανάσταση. Κατά τη γνώμη μου, η ελίτ στον καιρό της βιομηχανικής επανάστασης παίζανε διαφορετικό ρόλο δηλαδή στο πέρασμα από την αγροτική κοινωνία στην βιομηχανική κοινωνία. Σήμερα ο ρόλος του στην ψηφιακή επανάσταση είναι πιο περιορισμένος για τη συμβολή τους δηλαδή στην ανάπτυξη της ψηφιακής κοινωνίας. Επιμένω, ενιαία αγορά, ανταγωνιστική, ανοιχτή. Και επιμένω επίσης και στον ρόλο της έρευνας και της τεχνολογίας. Εγώ ορίζω 10 τομείς με συγκεκριμένους στόχους, ε, μεγάλους στόχους και ο καθένας από αυτούς ε, τους στόχους έχουμε τις, ε, τα policy goals και τα policy action πολιτικούς στόχους και πολιτικές δράσεις. Αυτές είναι οι προτάσεις μου. είναι κατεπίγουσα η εφαρμογή της νέας ε, νομοθεσίας για τις τηλεπικοινωνίες που εγκρίθηκε πρόσφατα. Και ή θα τροποποιήσουμε και θα συμπληρώσουμε έγκαιρα αυτή την νομοθεσία ή αλλιώς μιλάμε για να μιλάμε. Δηλαδή, αν δεν προχωρήσουμε και δεν έχουμε αλλαγές, τότε θα μείνουμε σε αυτά τα ποσοστά. Δηλαδή, κοιτάξτε, μόνο το 7% των συναλλαγών μέσω ίντερνετ είναι διασυνοριακές συναλλαγέ. Πρέπει λοιπόν να συμπληρώσουμε το πακέτο Telecom, είναι κατεπήγον πρέπει να γίνει έγκαιρα και ουσιαστικά σε όλες τις χώρες. Γι' αυτό ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τους Εθνικούς Ρυθμιστές, τον ΠΕΡΕΚ, ήδη έχει συσταθεί. και πρέπει να παίξει έναν σημαντικό ρόλο για να ρυθμίσει την κατάσταση και να παρεμβαίνει και στο μέλλον πιστεύω ότι είναι θεμελιώδες τόσο στη δική μας περίπτωση όσο και, στις, και, σε άλλες βέβαια να έχουμε παρακολούθηση αυτών των στόχων διότι αλλιώς θα έχουμε μία γνωμοδότηση παραπάνω και φτάνει πρέπει να έχουμε ένα μητρό ένα μητρό όπου θα καταγράφονται τα πεπραγμένα πρέπει να καταγράφονται οι πρόοδοι σε όλους τους τομείς Και τελειώς να καταλήξουμε πουθενά και τίποτα άλλο. Και να πω και κάτι άλλο ότι η παρέμβαση των συναδέλφων αυτή η ψηφιακή ατζέντα δεν έχει ως στόχο να ξανανοίξει το πακέτο για τις τηλεπικοινωνίες και να ερμηνεύσει το πακέτο της Τελεκόμ. Ε, τροπολογίες που εγώ τις γνωρίζω πολύ καλά, εντάξει, σύμφωνοι. Υπάρχει πειρασμός βέβαια. Δεν έχει νόημα λοιπόν να ανοίξουμε, είπαμε, το πακέτο. Εγώ Προτείνω λοιπόν αυτό το έγγραφο με αυτές τις προτάσεις ε, που ερμηνεύουν αν θέλετε τις θεματικές του πακέτου δεν θέλω να ξανανοίξω το πακέτο το δηλώνω αυτό θα τα ξαναπώ στο τέλος σας ευχαριστώ Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη σημαντική αυτή εισαγωγή και παρουσίαση για να ξέρουμε τι θα αποτελέσει και το περιεχόμενο της συζήτησης. Έχω δέκα συναδέλφους που έχουν ζητήσει το λόγο να παρακαλέσω τους συναδέλφους να περιοριστούν λίγο χρονικά και θα βάλουμε και το ρολόι. Ο κύριος Βικμαρκ έχει το λόγο καταρχάς. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγητρία καταρχάς που μας εξήγησε και μου έκανε την εισαγωγή για τη συζήτηση αυτή για τη νέα ψηφιακή ατζέντα, γιατί πρόκειται για ένα από τα πιο βασικά πράγματα που μας απασχολούν. Θα ήθελα να παρουσιάσω κάποιες διαστάσεις που είναι σημαντικές, θεωρώ, για το επόμενο βήμα. Καταρχάς, οι βασικές αλλαγές που γίνονται σε παγκόσμιο επίπεδο μετά την κρίση γιατί φυσικά πριν ήταν η Ευρώπη και η ΕΠΑ οι οποίες από αν θέλετε ήταν ε, στην κορυφή των ψηφιακής ε, ε, προόδου. Η Ευρώπη ήταν παγκόσμιο φορέας, αλλά τώρα βλέπουμε ότι τα αριθμητικά στοιχεία καταδεικνύουν ότι έχουν αλλάξει πλέον τα πράγματα. Η Κίνα και η Ινδία θα καταστούν όλο και πιο δυνατές αγορές. Και βλέπουμε ήδη σήμερα ότι οι βασικοί φορείς τελεκόμ, επικοινωνιών είναι ε, από κινέζικη, κινέζικης προέλευσης. Ένας μόνο είναι Ευρωπαίος. Και όλα αυτά φυσικά θα θέτουν τις βάσεις για τη μετέπειτα εξέλιξη της, ε, του κλάδου. Και νομίζω λοιπόν ότι στο πλαίσιο αυτό να έχουμε υπόψη ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση ο μεγαλύτερος βαθμός εξέλιξη και, και διείσδυσης των νέων τεχνολογιών είναι κυρίως στα τμήματα εκείνα της Ένωσης, όπου υπάρχει πιο ανοιχτός χαρακτήρας για νέες εισόδους εταιριών και πιο πολύ ανταγωνισμό. Αυτό είναι σημαντικό να το έχουμε υπόψη. Όπως υπογράμμισε και η συγγήτρια, υπάρχει ανάγκη να εφαρμοστεί το πακέτο τηλεπικοινωνιών. Θα είναι βασική ε, και ζωτική σημασία σε αυτό για το μέλλον. Τρία στοιχεία θέλω να θίξω επιπρόσθετα, αν θέλετε, πέρα από αυτά που έχουν ήδη ακουστεί. Θεωρώ ότι τρία σημεία θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε με μεγαλύτερη, ε, μεγαλύτερο στένο. Το ψηφιακό αυτό, αν θέλετε, ε, το ψηφιακά προϊόντα, τα οποία θα πρέπει να είναι τα οποία θα πρέπει να ασκήσουμε στα κράτη-μέλη, προκειμένου να γίνει η καλύτερη δυνατή χρήση των ψηφιακών αυτών προϊόντων για να υπάρχουν νέες λύσεις, νέες υπηρεσίες σε ό,τι αφορά το φάσμα. Αυτό καταρχάς. Καταρχάς, κατά δεύτερον, το ηλεκτρονικό εμπόριο. Θα πρέπει να συνδέσουμε την ψηφιακή ανάπτυξη με τον υπόλοιπο κόσμο. Νομίζω ότι μία μεταρρύθμιση που θα πρέπει να γίνει είναι να υπάρχουν ε, σημεία επαφής σε όλα τα κράτη-μέλη για το ΦΠΑ για να είναι πολύ πιο ε, εύκολες και γρήγορες οι ψηφιακές συναλλαγές και για τον καταναλωτή αλλά και για τις εταιρείες. Να μην υπάρχουν πλέον τα γραφειοκρατικά εμπόδια που υπάρχουν σήμερα για την ηλεκτρονικό εμπόριο. Είναι απλή αυτή η μεταρρύθμιση ίσως, αλλά θα πρέπει να μπει στην ημερήσια διάταξη για είναι συνάδεια, αν θέλετε, η ψηφιακή πρόοδος με την πρόοδο της ενιαίας αγοράς. Κατά τρίτον, σε ό,τι αφορά τις επενδύσεις στις νέες τεχνολογίες, πιστεύω ότι θα χρησιμοποιήσουμε τις επενδύσεις της αγοράς ε, όσο το δυνατόν καλύτερα να διασφαλίσουμε ιδιωτικές και δημόσιες επενδύσεις οι οποίες δεν θα γινόντουσαν υπό άλλες συνθήκες. Θα πρέπει να υπάρχει λοιπόν ε, μεγάλη συμμετοχή στην ψηφιακή αγορά. Εκ παραλίλου όμως να κάνουμε και κάτι άλλο. Να διασφαλίσουμε ότι όταν επενδύουμε πάντα να επενδύουμε στην πιο ε, κορυφαία τεχνολογία, στην πιο σύγχρονη τεχνολογία. Αυτό σημαίνει από φιλοσοφικής άποψης για την πρόοδο της ψηφιακής ε, αγοράς, θα πρέπει να υπάρχει ευρεία χρήση, ευρεία αξιοποίηση των ψηφιακών δυνατοτήτων και θα πρέπει επίσης να συγκεντρώσουμε την ελίτ. Γιατί αν δεν ε, είμαστε πιο γρήγοροι στην εξέλιξή μας από άλλες περιφέρειες, θα μας κερδίσουν αν θέλετε στον ανταγωνισμό επειδή είναι πιο μεγάλες αριθμητικά. Ευχαριστώ και πάλι την εισηγήτρια για τις συζητήσεις που κάναμε για να ενισχύσουμε αυτή την ευρωπαϊκή ψηφιακή ατζέντα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Τσουκαλάς. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω την ερήτημη κυρία Πιλάρντε Καστίγιο για την πολύ ευχάριστη έκπληξη που απετέλεσε για μένα το κείμενό της, αρχίζοντας από την αιτιολογική έκθεση και καταλήγοντας στο σχέδιο ψηφίσματος. Ο κύριος Χέκμακ με απίλαξε με τις εύστοχες παρατηρήσεις μου της υποχρέωσης να αναφερθώ στα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα που είπε. Θα αντιμετωπίσω το κείμενο της κυρίας Πλέρ Δεκαστήγιο ως ένα κείμενο που είμαι βέβαιος ότι στους στην αγορά αλλά και στους ακαδημαϊκούς κύκλους θα γίνει ένα best seller. Έχει όλα τα προσόντα, έχει την, το απαραίτητο μίξ ρεαλισμού και ιδεαλισμού, διαθέτει όραμα, αποστολή και στόχους, χαράσει στρατηγική και πολιτική, θέτει στη διάθεσή μας τις τάξεις και τις τάξεις των εργαλείων που χρειάζονται, επισημαίνει την ανάγκη ύπαρξης ενός προγράμματος δράσης, καθώς επίσης επικεντρώνει την όλη του φιλοσοφία στον άνθρωπο. Μιλώντας για τον άνθρωπο, τώρα στους καιρούς μας, συνηθίζουμε να τον βλέπουμε τον άνθρωπο είτε ως μια παραγωγική μηχανή, είτε ως ένα σύνολο δικαιωμάτων. Η εποχή μας, με τη βοήθεια της ψηφιακής εποχής, έχει μετατοπίσει, όπως είπε και η κυρία Καστίγιο, τα φυσικά πλεονεκτήματα της παραγωγής από τα μηχανήματα ή τους φυσικούς πόρους ή το κόστος εργασίας στο κατακεφαλή περιεχόμενο πολιτιστικό και επιστημονικό του ανθρώπου. Αυτό μετατρέπει την υποχρέωση της πολιτείας να καθιστά τους πολίτες ικανούς να έχουν μια ζωή με νόημα, ταυτόχρονα και ένα προαπαιτούμενο για παραγωγή, η οποία παραγωγή μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο από ανθρώπους που έχουν αυτό το παράλληλο μίξ. Ζούμε σε μια εποχή όπου ο άνθρωπος είναι το ίδιο αγράμματος όταν δεν ξέρει το δεύτερο θερμοδυναμικό αξίωμα ή δεν έχει διαβάσει Τσέχοφ ή Θερβάντες. Η πραγματική ερμηνεία του εξωτερικού αντικειμενικού κόσμου έχει την απέτηση για την ακρίβεια της ερμηνείας της, της κατάρτισης του ενός ορίου κατάρτισης, κάτω από το οποίο το όραμα που έχει ο σύγχρονος άνθρωπος για μια κοινωνία συνεκτική περί της αξίες και σε μια ατομική ζωή με νόημα δεν μπορεί να επιτευχθεί. Με αυτή την έννοια το κείμενο της κυρίας Ντεκαστήγιο είμαι βέβαιος ότι θα τραβήξει την προσοχή όλων των συναδέλφων είτε ανήκουν είτε δεν ανήκουν σε αυτή την ε, Επιτροπή ε, και είμαι βέβαιος ότι όλοι θα προσπαθήσουμε να δώσουμε και τη δική μας συμβολή. Ε, παραδείγματι, μιλώντας για τον άνθρωπο, είναι προφανές ότι στην παραγωγή οι νέοι άνθρωποι που θα μείνουν αποκλεισμένοι από αυτές τις δεξιότητες θα είναι σε χειρότερη θέση από τους ηλικιωμένους ανθρώπους που σήμερα δεν τις έχουν. Γιατί εκείνοι στις παραγωγικές ε, δυνατότητές τους ε, δεν θα έχουν τα απαραίτητα μέσα παραγωγής όπως αυτή σήμερα διαμορφώνεται. Και θα έχουμε και πάλι μια, ε, ένα διαχωρισμό αν η Ευρώπη, αν τα κράτη-μέλη δεν στήσουν την προσοχή τους με τη σοβαρότητα που τη στείλουν άλλα κράτη. Για παράδειγμα να σας υπενθυμίσω την αμφιλεγόμενη Τουρκία η οποία με πρόσφατο νόμο αποδίδει διευθύνσεις IP με την γέννηση κάθε πολίτη της, όπως ακριβώς κάνει από την εποχή Κλίντον η Αμερική για τους Αμερικάνους πολίτες. Τέλος, πραγματικά χρειάζεται η Ευρώπη μεγαλύτερη ταχύτητα και τόλμη. Για παράδειγμα, εάν δεν βιαστούμε για την Ευρωπαϊκή, το Google θα την καταστήσει άχρηστη. Γιατί απλούστατα εμείς διστάζουμε και ένα πλούτο 27 κρατών μελών ή μιας ευρωπαϊκής παράδοσης και μιας παράδοσης της Ευρώπης 400 ετών σε πνεύμα επιστήμη και τέχνες δεν μπορεί να έχει την ψηφιακή της απεικόνηση με την ταχύτητα και τον πλούτο που χρειάζεται. Από αυτή την έννοια την κυρία Καστίγιο να ευχαριστήσω και να επισημάνω το πολύ καλό για μένα έργο που είδα. Σε ευχαριστώ πολύ. Äh, Ο συνάδελφος Καλφίν, σκιώδης εισηγητής. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα να συγχαρώ την κυρία Δελκαστηγιό για το σχέδιο έκθεσης το οποίο αποτυπώνει σε μεγάλο βαθμό, θεωρώ, τη σημασία της ε, εξέλιξης των ψηφιακών τεχνολογιών. Επίσης, θέτει συγκεκριμένους στόχους, συγκεκριμένες φιλοδοξίες για τα επόμενα πέντε έτη και είναι πάρα πολύ σημαντικό οι Ευρωπαίοι πολίτες να τοποθετηθούν στο, στον πυρήνα της εξέλιξης των τεχνολογιών αυτών και φαντάζομαι ότι ο νέος ο επιτρεπός, ο οποίος ήταν αποκλειστικά υπεύθυνο με την ψηφιακή ατζέντα, είναι επιτροπός, θα μπορέσει να πετύχει συγκεκριμένες νίκες σε ό,τι αφορά την ψηφιακή τεχνολογία. Θα ήθελα να υποστηρίξω τώρα κάποια βασικά στοιχεία αναφορικά με την εκθέση της κυρίας Τελκαστήγιο. Καταρχάς, σε ό,τι αφορά την εισαγωγή συγκεκριμένων παραμέτρων για την πρόωθηση των ψηφιακών τεχνολογιών. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με καλύτερο περιβάλλον ανταγωνισμού. Γιατί είναι σαφέ όπου υπάρχει πιο πολύ ανταγωνισμός, οι πολίτες έχουν μεγαλύτερη, γρηγορότερη πρόσβαση και φθηνότερη πρόσβαση στο ίντερνετ. Κατά δεύτερον, θα πρέπει να δημιουργηθούν φιλοδοξίε για να χρησιμοποιηθούν πιο πολλέ. Ε, υπηρεσίες μέσω του διαδικτύου και θα πρέπει προς το σκοπό αυτό να κοιτάξουμε πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε μια ενιαία, πραγματικά ενιαία αγορά προϊόντων και υπηρεσιών στο διαδικτύο και επίσης θα πρέπει να εκπαιδεύσουμε τους πολίτες, όλους τους πολίτες για τη χρήση της ε, ψηφιακής τεχνολογίας. Υπάρχουν κάποια λοιπόν στοιχεία που θα ήθελα να υπογραμμίσω θεωρώ ότι το Κοινοβούλιο θα μπορέσει να συμμετάσχει στα στοιχεία αυτά. Καταρχάς, οι ψηφιακές τεχνολογίες έχουν νόημα μόνο αν διασφαλίζουν καλύτερη ποιότητα ζωής, καλύτερη ποιότητα δουλειάς για τους Ευρωπαίους πολίτες. Και εδώ βασικό είναι, επειδή όλοι βλέπουμε τις επαναστατικές αυτές αλλαγές στην καθημερινή μας ζωή, χάρη στην τεχνολογία, σημαντικό είναι να μην επιτρέψουμε να δημιουργηθούν ε, χάσματα, να μην δημιουργηθεί ψηφιακό χάσμα. Και γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να σκεφτούμε ιδιαίτερα την αρχή της αλληλεγγύης στο πλαίσιο της ε, κοινωνίας, της ψηφιακής πληροφορίας. Κατά δεύτερον, να ρωτήσω, γιατί ύστερε η Ευρώπη σε ό,τι αφορά τα νέα προϊόντα και τις νέες υπηρεσίες ε, στην ψηφιακή τεχνολογία. βλέπουμε ότι η ευρωπαϊκή αγορά είναι κατακαιρματισμένη. Ωστόσο δεν φταίει μόνο αυτό. Είναι απαραίτητο να υπάρχουν πιο πολλά κίνητρα και για τα πανεπιστήμια και για τα ερευνητικά κέντρα και για τις εταιρείε προκειμένου να συνεργαστούν για τη δημιουργία νέων ευρωπαϊκών αγορών, τα οποία θα προωθηθούν καταρχάς στις ευρωπαϊκές αγορές. Κατά τρίτον, όταν μιλάμε για νέα προϊόντα και για νέες τεχνολογίες, αντιμετωπίζουμε αναπόφευκτα το πρόβλημα του περιεχομένου του διαδικτύου είναι σαφές ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει περιθώριο να αναβάλει τη συζήτηση αυτή. Θα πρέπει να βρει μακροπρόθεσμες λύσεις αποδεκτές και από την κοινωνία που θα συμβάλλουν στη δημιουργία νέων προϊόντων στο διαδικτύο. Δεν μπορούμε να περιορίζουμε την ανάπτυξη του διαδικτύου και θα πρέπει να δώσουμε και σαφείς απαντήσεις σε ό,τι αφορά τη ρύθμιση του περιεχομένου. Αυτό σημαίνει ότι τα κοινωνικά πρότυπα θα πρέπει να προσαρμοστούν στο νέο ψηφιακό περιβάλλον και μάλιστα όσο το γρηγορότερο δυνατόν. Τέλος, τίθεται και το θέμα της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο δεν επαρκεί η επικύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης. Θα πρέπει να επιτύξει μεγαλύτερη ε, δραστηριότητα η Ευρωπαϊκή Ένωση σε ό,τι αφορά την καταπολέμηση του κυβερνού κλίματος. Επίσης, θα πρέπει να υπάρξει και ευρωπαϊκός συντονισμός. Δεν πρόκειται να επισέλθω σε λεπτομέρειε, αλλά η ψηφιακή Ευρώπη δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί χωρίς πραγματικά ασφαλή κυβερνοχώρο. Το θέμα αυτό θα μπορούσαμε να το τονίσουμε λίγο πιο έντονα στην έκθεση. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος, η συνάδελφος Βαλεάν. thank you, Ευχαριστώ, Πρόεδρο. Θα ήθελα καταρχά να ευχαριστήσω την κυρία Τελφά στην Κλουβιέρα για την εκκλησία τη Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα, ήταν πολύ καλέ οι ιδέε και οι οι έννοιε τι οποίε έχει αναπτύξει, συμφωνώ με του τομεί δράση και πολιτική που έχει ε, προβάλλει στην εκθεσή της και την ανάγκη να αναπτυχθεί η καλύτερη η ψηφιακή κοινωνία, η, ιδιαίτερα με την ευρυζωτικότητα και τη δυνατότητα για τον πολίτη να συμμετέχει σε μια ε, ανοιχτή κοινωνία ψηφιακή που θα επιτρέψει τον πολίτη να έχει πλήρη αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στα προσεχή χρόνια. Και επίσης συμφωνώ ότι θα πρέπει να έχουμε μια συνεκτική στάση και όσο το δυνατόν πιο πολύ ε, αντίκτυπο στις προσπαθίες μας. Δεν θα πρέπει ωστόσο και να επαναπροσδιορίσουμε έννοιες ήδη εδρεωμένες, εδρεωμένες όπως ψηφιακή διακυβέρνηση. Και θα ήθελα να διευκρινίσουμε το εξή. Το 2015 είναι ε, ρεαλιστικό στόχο άραγε με δεδομένη και τη στρατηγική 20-20-20 ε, για την ε, ενιαία αγορά online. Και μέσα από τη διαδικασία, την ολοκλήρωση διαδικασία για τη λήψη αποφάσεων και την ε, διαδικασία για, τη λήψη, για την έγκριση των κανονισμών και την εφαρμογή της όσο έχουμε ξεπεράσει το 2015 πολύ γρήγορα. Με το 2020 λοιπόν και την ενδιάμεση αναθεώρηση θα, θα μπορούσαμε να αλλάξουμε τις προθεσμίες. Δηλαδή θα μπορούσαμε να πούμε το 2015 είναι για την ενδιάμεση αναθεώρηση. Επίσης για μια πρόσθετη οικουμενική υπηρεσία για την ευρυζωνικότητα. Αυτή η απέτηση νομίζω θα πρέπει να αναθεωρηθεί, να έχουμε μια πιο δυναμική προσέγγιση, μια προσέγγιση προσαρμοσμένη στην συνθήκε αγορά των τηλεπικοινωνιών. Ε, παραδείγματι αποτελεσματική ανταγωνιστικότητα ω προ την υπηρεσία, ε, αποτελεσματική λειτουργία τη αγορά ε, και όχι ε, επιδοτήσει ή ενισχύσει για επενδύσει. Και Πιστεύω ότι χρειάζεται περισσότερη ανταγωνιστικότητα στην αγορά ε, και στη σταθερή τηλεφωνία για να μην διατηρούν οι παλαιές εταιρείε, οι πρώην μονοπωλιακές εταιρείε όλα τα πλεονεκτήματα. Ιδιαίτερα δε ως προς τους συγκεκριμένους κανονισμούς κοινωνιών που αναφέρεται στην παράγραφο αριθμών 7 που θα πρέπει εκ των προτέρων να καταργηθούν δεν μπορώ να συμφωνήσω. Πιστεύω ότι το πλαίσιο της Επιτροπής είναι κατάλληλο για τις επιχειρήσεις και είναι αυτό το οποίο προσφέρει τα καλύτερα αποτελέσματα και, συμφε... και πλεονεκτήματα για τον καταναλωτή. Θα πρέπει οι ειδικοί κανονισμοί να καταργούνται μόνο όταν έχει αποδεδειγμένα εξασφαλιστεί αποτελεσματικός ανταγωνισμός. Και έχω πρόσθετε ιδέε επίση να προσθέσω, τι οποίε ενδεχομένω να θέλετε να λάβετε υπόψη στην ε, έκθεσή σα. Η ψηφιακή ατζέντα θα πρέπει να προάγει μακροπρόθεσμο και βιώσιμο ανταγωνισμό μεταξύ παραγόντων των υποδομών, φορέων των υποδομών ε, και θα πρέπει να διατηρηθούν οι, ε, τα κίνητρα για περισσότερε επενδύσει και τώρα και στο μέλλον, καλύτερες επενδύσεις και τώρα και στο μέλλον, με δεδομένο ότι θέλουμε να έχουμε υποδομές ανοιχτέ, υποδομές που ενισχύουν και διευκολύνουν την καινοτομία και τη διαφοροποίηση για το των καταναλωτών. Και επίσης τηλεφωνία είναι κατακαιρματισμένη η αγορά, ε, δεν υπάρχουν απαραίτητα πάντοτε τα κίνητρα για περισσότερε επενδύσεις ή διαφοροποιημένες επενδύσεις. Χρειάζεται λοιπόν να ενισχύσουμε την έννοια της ευρυζωνικότητας για καλύτερες και ταχύτερες υπηρεσίες και τόσο η διαφοροποιημενες επενδυσεις χρειαζεται λοιπον να ενισχυσουμε την εννοια τη ευρυζωνικοτητας για καλυτερες και ταχυτερες υπηρεσιες και τοσο η κατανομη του ψηφιακού μερίσματος όσο και η βελτίωση των τιμών για την καταναλωτή θα πρέπει να διευκολύνουν τον, τον χώρο της ε, τηλεφωνία στην παράγραφο 4 θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι δεν θα πρέπει να ε, δώσουμε έμφαση στην ε, τεχνολογία του 3G αλλά περισσότερο ε, στην ευρυζωνικότητα και στην καλύτερη κατανομή του ψηφιακού μερίσματος. Η αγορά επιπλέον δεν θα πρέπει να περιοριστεί μόνο ή να θεωρηθεί μόνο μια αγορά λιανική που στοχεύει μόνο στον ιδιώτη καταναλωτή. Πρέπει να λάβουμε υπόψη και τι ανάγκε των επιχειρήσεων και ιδιαίτερα στην Ευρώπη, τι μικρομεσαίε, αλλά και τι ε, πολυεθνικέ που θα πρέπει να είναι σε θέση να προσφέρουν τεχνολογικά προϊόντα, τι νέε τεχνολογίε, σε ανταγωνιστικέ τιμέ. Οι εταιρείε σε ένα κράτο μέλο θα πρέπει να έχουν την ίδια ε, ισότιμη δυνατότητα πρόσβαση στο δίκτυο των τηλεπικοινωνιών και προβλέπεται ότι οι επιχειρήσει θα είναι εκείνε οι οποίε θα διαδραματίσουν τον κύριο ρόλο προ την προγωγή διαφορετικών διαφορετικών πλατφορμών και υπηρεσιών όπως cloud computing, smart grids ή, ή ηλεκτρονικής υγείας. Ευχαριστώ. Είχα και άλλα να πω, Πρόεδρε, αλλά ευχαριστώ, δεν χρειάζεται. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος, ο τους δυο Τώρα ο κύριος Λάμπερτς έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εδώ είμαστε στην Επιτροπή Βιομηχανίας. Θα ήθελα λοιπόν να κοιτάξω μια πιο βιομηχανική σκοπιά στην υπόθεση αυτή. Αγορά. Αγορά τι σημαίνει. Σημαίνει υποδομές, και εδώ θα έλεγα να μην ε, επαναπαυόμεθα στις δάφνες μας, διότι η τεχνολογία έχει φέρει την Ευρώπη στην κατώτερη δυνατή θέση. Μπορεί να έχουμε υποδομές ε, και παρόχους που χρησιμοποιούν κάποια υποδομή, αλλά δεν υπάρχει τελευταία τεχνολογία. Ο κύριο Κολασάντη διαφωνεί, ίσω ναι, αλλά δεν είμαστε, οι Ευρωπαίοι δεν είναι οι ηγετικές επιχειρήσεις. Μπορείτε να μου πείτε ότι στην κινητή τηλεφωνία η Nokia καινοτομή κτλ. Αλλά όχι, δεν είναι ευρωπαϊκή τεχνολογία εχμή αυτή τη στιγμή. Δεύτερον, στις εφαρμογές, εκεί που ουσιαστικά βγαίνουν και τα πολλά κέρδη το λογισμικό που παράγεται στον πλανήτη μας πάλι δεν προέρχεται κατά κύριο λόγο από την Ευρώπη. Αντί λοιπόν να επαναπαυόμεθα θα πρέπει να κινητοποιηθούμε για να κερδίσουμε μεγαλύτερο μερίδιο στις αγορές αυτές. Και ευχαριστώ πολύ την Πιλάρ που μας έδωσε το αρχικό αυτό σχέδιο και τις προσπάθειές της, αλλά θέλω να σημειώσω ότι δεν είναι για μένα τόσο επίγουσα αυτή η προοπτική. Δεύτερον, πού πάει η αγορά. Αν δούμε την ε, τεχνολογία της πληροφορίας, αρχικά στόχος ήταν η παραγωγικότητα των ανθρωπίνων πόρων. Αυτό περισσότερο έχει εξασφαλίσει η πληροφορική τις τελευταίες δεκαετίες. Η αγορά όμως σημαίνει τώρα πια ε, και ενεργειακή παραγωγικότητα και παραγωγικότητα πόρων που πάλι χάρη στις εφαρμογές θα, το, θα εξασφαλίσουμε και όχι χάρη στο υλικό, το hardware. Ο χώρος για το hardware έχει χαθεί, ας τον αφήσουμε. Πολιτισμός, ε, διάδοση πολιτισμού, νέες δυνατότητες και όπως είπε εκεί στην Αρφή η ηλεκτρονική υγεία είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα. Σε μια γυράσκουσα κοινωνία είναι σημαντικό να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε την παραμονή των ηλικιωμένων στο σπίτι τους, ε, στην κοινωνία όπου ζουν, στη γειτονιά τους, αντί να τους παρκάρουμε σε κάποιο ειδικευμένο γεροκομείο οίκο ε, αυτό λοιπόν που θα κερδίσει την αγορά είναι οι εφαρμογές και εδώ ακριβώς βλέπω την βιομηχανική σκοπιά. Ε, η Ευρώπη για να μπορέσει να ηγηθεί δεν μπορώ να πω γιατί αργού, αργήσαμε να ξεκινήσουμε αλλά για να έχουμε μια καλή παρουσία περιπτώσει πρέπει να επιταχύνουμε τους ρυθμούς μας και άκουσα να μιλούν για ανταγωνισμό και ανοιχτή αγορά κτλ. Οι συνάδελφοι, ναι συμφωνώ Όντω. Αλλά το να έχουμε μόνο μια ανοιχτή αγορά χωρίς κίνητρα, χωρίς στόχους, χωρίς δημόσιες επενδύσεις ως προς την επιτάχυνση της έρευνας που θα μας επέτρεπε να κερδίσουμε το χαμένο έδαφος, δεν θα μας φέρει κανένα αποτέλεσμα. και θα έλεγα ότι μπορούμε να κάνουμε και τη σύγκριση μεταξύ στρατηγικής Λισαβόνας και της στρατηγικής του 2010. Αν δούμε την ουσία και τα επιτεύγματα, καταλαβαίνουμε τι άλλο έχουμε να, τι, πόσο πολλά μένουν να γίνουν. Επίσης τα δικαιώματα των χρηστών Προσπαθήσαμε με την τροπολογία 138 να αξιοποιήσουμε κάθε τύπου νομοθεσία, είτε, για τη βιο... είτε νομοθεσία σχετική με τι αγορέ, είτε με τη βιομηχανία κτλ. Και προσπαθούμε να προσδιορίσουμε τι είναι, ποια είναι τα δικαιώματα του καταναλωτή, του χρήστη δηλαδή ίντερνετ εν προκειμένου στην Ευρώπη. Και ε, χρειάζεται πιστεύω ένας χάρτης δικαιωμάτων των καταναλωτών χρηστών του ίντερνετ του διαδικτύου που θα προσδιορίζει και τα δικαιώματα στην πρόσβαση βεβαίως και το δικαίωμα στην ασφάλεια και υπενθυμίζω τα όσα είπα για την ασφάλεια των δικτύων, αλλά και το δικαίωμα στην προστασία του ιδιωτικού βίου. Παράδειγμα, εάν θέλουμε να έχουμε μια κοινωνία χαμηλής ενέργειας, χαμηλής κατανάλωσης ε, άνθρακα, μιλάμε συνήθως ε, για ευφυή κινητικότητα, ε, δηλαδή κατά την ανάγκη ε, πληρωμή. Πληρώνω ανάλογα με τα μέσα ε, μαζικών μεταφορών που χρησιμοποιώ. Αυτό όμω σημαίνει ταυτόχρονα και παρακολούθηση από κάποιο κέντρο του που βρισκόμαστε. Δηλαδή κάποιο θα γνωρίζει ανά πάσα στιγμή που βρισκόμαστε. Τέλο πάντων, είναι υπερβολική αυτή η ιδέα, αλλά αυτή είναι η ιδέα και έτσι σε μια αντίστοιχη περίπτωση θέλουμε να έχουμε επαρκή εγγυήσει για την προστασία του ιδιωτικού βίου. Φυσικά αυτό θα πρέπει να απασχολεί στην Επιτροπή Μηχανία, αλλά πρέπει να το αναλάβει η ΛΥΜΠΕ είτε κάποια άλλη αντίστοιχη επιτροπή. Και οι στόχοι θα πρέπει να ορίζουμε βεβαίω ότι πρέπει να γίνει, αλλά όχι αποκλειστικά και μόνο στον χώρο τη ε, πληροφορική. Ο στόχο ε, φερειπίν τη μείωση των εκπομπών. Αν δεν είναι φιλόδοξο, αν δεν είναι φιλόδοξοι όλοι μα οι στόχοι, δεν θα βοηθήσουν την ευρωπαϊκή βιομηχανία στο να αναλάβει τα ενία ε, το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο που βρίσκεται υπό εκτέλεση, το 8ο πρόγραμμα πλαίσιο που ε, προχωράει σε ε, εφαρμογή σιγά σιγά. Όλα αυτά πρέπει να έχουν αυτές τις διαστάσεις της νέας τεχνολογίας και της πληροφορικής. Βεβαίως υπάρχουν πολλά καλά στοιχεία στην έκθεση πρέπει να πω, αλλά, αλλά δεν συμφωνώ ότι θα αποτελέσει ένα σημείο αναφοράς για χρήση από, την, από τον νομοθέτη, από τις ε, επιχειρήσεις κτλ. Δεν βλέπω αρκετά σαφείς όρους. Πρέπει να είναι πιο σαφές το κείμενο, πρέπει να είναι πιο φιλόδοξο και συγκεκριμένο. Και βέβαια το 2015 παρά είναι φιλόδοξο και δεν θα μπορέσει να επιτρέψει στην Ευρώπη να προετοιμαστεί επαρκώ για να αναλάβει τα, τα ίνια. Και παραλαμβάνω, δεν πρέπει να επαναπαυόμεθα. Ναι, υπάρχουν κάποιες ε, Επιχειρήσει όπω η Nokia ή η SAP που πάνε καλά, αλλά δεν αρκούν αυτά για να αναλάβει η Ευρώπη ηγετικό ρόλο στη παγκόσμια σκηνή. Πρέπει να προχωρήσουμε ακόμα καλύτερα. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα ακούσαμε όλου και οδηγητέ, αγαπητοί συνάδελφοι. Αν παίρνει ο καθένα 6 6-7 λεπτά με την ομιλία, δεν θα προλάβουμε να τελειώσουμε. Παρακαλώ, το πολύ πολύ στα 2 λεπτά. Ε, για να ακούσουμε λοιπόν τους επόμενους ομιλητές. Πρωτικό. Um, ε, κυρία Τικάουν, ευχαριστώ πρόεδρε, αλλά η κυρία Φιγκαρίδο είναι η σκιώδη συγγετριά. Ίσως να της δώσουμε το λόγο πρώτης. Μα ναι, ναι, ναι, εννοείται, εννοείται, λέει ο πρόεδρος. Έχετε το λόγο κυρία Φιγκαρίδο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, πράγματι εδώ εκπροσωπώ εγώ την ομάδα της ΓΚΟΕ και θα παρακολουθήσω εγώ αυτήν την έκθεση. Θα ήθελα σύντομα να υπογραμμίσω, δεν θα είμαι μακροσκελής, αλλά θα υπογραμμίσω τρία ζητήματα. Εγώ πιστεύω ότι η έκθεση που παρουσίασε η συνάδελφος είναι πολύ ισορροπημένη Βέβαια, κατά τη γνώμη μου, μπορούμε να βελτιώσουμε τις διάφορες προτάσεις ε, που υποβλήθηκαν και που είναι σημαντικές για να αποφύγουμε να έχουμε εκ νέου κοινωνικό αποκλεισμό από την ψηφιακή εξέλιξη. Και θέλω να επιστήσω την προσοχή σας αυτό το ευρωπαϊκό έτος για την καταπολέμηση της φτώχειας. Πρέπει να έχουμε προτάσεις οι οποίες θα ελκύουν το ενδιαφέρον για τα υφιστάμενα προβλήματα και οι προτάσεις επίσης που θα υποβληθούν δεν θα πρέπει να επιφέρουν παραπάνω ανισορροπία, παραπάνω αποκλεισμό, παραπάνω διαφορές και διακρίσεις μεταξύ των κοινωνικών στρωμάτων, κυρίως αυτών που δεν έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης. Εγώ ε, αναλογίζομαι πόσο σημαντικό μπορεί να είναι ο ψηφιακός τομέας για να βοηθήσει ορισμένα κοινωνικά στρώματα, ας πούμε τους αναπήρους. Για τους αναπήρους η ψηφιακή εξέλιξη μπορεί να αποτελέσει σημαντικό μέσο κοινωνικής ένταξης Εγώ θεωρώ ότι οι δημόσιες επενδύσεις είναι σημαντικές σε αυτόν τον τομέα. Αλλά θα πρέπει να δούμε πώς θα αναπτύξουμε και την αρχή της αλληλεγγύης ούτως ώστε να μην ενταθούν οι ανισότητες Εσείς ε, κάνετε ορισμένες νήξεις στην έκθεσή σας, δηλαδή από τώρα μέχρι το 2015, να μην μεγαλώσουμε το χάσμα μεταξύ των λαών, των χωρών, των περιφερειών. Επίσης οι συνάδελφοι μίλησαν για την προστασία του ιδιωτικού βίου, επέστησαν την προσοχή μας ε, για την cyber ε, ε, εγκληματικότητα, αλλά όλα αυτά ισχύουν όχι μόνο για τον ψηφιακό τομέα, ισχύουν και για το εμπόριο, ισχύουν ε, και για το ίντερνετ σήμερα όπου χρειάζεται δηλαδή να έχουμε νομοθεσίες τέτοιες που να μην οδηγούν σε αποκλεισμό ε, μικροεπιχειρήσεων, καταναλωτών κλπ που μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτές τις υπηρεσίες. Πρέπει λοιπόν όλοι να έχουν πρόσβαση σε αυτόν τον πλούτο του ψηφιακού κόσμου. Αλλά προσοχή διότι μπορούν να αυξηθούν οι κοινωνικές ανισότητες και έχουμε σε αυτόν τον τομέα ακόμη μερικές προτάσεις να υποβάλουμε. Κύριε Τιτσάου, Πρόεδρε, ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω, να συγχαρώ την ε, εισηγήτρια και να ζητήσω μια ε, δυνατότητα για από κοινού αναλογισμό του τι έχουμε κάνει για το 2010, πού βρισκόμεθα, ποιοι είναι οι λόγοι για τους οποίους οι στόχοι που είχαμε ορίσει δεν επετεύχθησαν 100%. Φερρυπίν, γνωρίζουμε ότι το Ευρωπαϊκό Σχέδιο Οικονομικής Ανάκαμψης κόστισε μερικά δισεκατομμύρια δολάρια. Και φτάσαμε στο τέλος ε, του 2010 με κάλυψη 5% μόνο ευρυζωνικότητα ε, για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά. Ε, ας δούμε λοιπόν τι κάναμε, τι δεν έχει γίνει και τι προτείνουμε για το 2015. Ε, δεύτερον, πιστεύω ότι η ηλεκτρονική διακυβέρνηση είναι πολύ σημαντική και ιδιαίτερα εννοώ τη σχέση μεταξύ αρχών και πολιτών, την επικοινωνία αρχών με τους πολίτες, μάλλον πολιτών με τις αρχές, ε, με ηλεκτρονικό τρόπο. Είχαμε πολλές ε, προόδους ως προς τις ηλεκτρονικές πληρωμές και την ηλεκτρονική υγεία, το e-health, Ξέρετε, έγιναν πολλές προσπάθειες και για την ηλεκτρονική τιμολόγηση, τα ηλεκτρονικά τιμολόγια ή invoice, αλλά από όλη την οδηγία για τις υπηρεσίες ε, υπάρχει ακόμη η προϋπόθεση το 2012 να μπορούν οι πάροχοι των υπηρεσιών σε όλη την Ευρώπη να είναι σε θέση να παρέχουν τις υπηρεσίες τους ηλεκτρονικώς, πράγμα μας το οποίο δεν έχει ακόμη επιτευχθεί. Φερρυπίν ε, δεν μπορεί κάποιος από την Πορτογαλία να συμμετάσχει σε ένα σεμινάριο στην ε, Γαλλία. Χρειάζεται να έχει ε, την ηλεκτρονική υπογραφή για την οποία πρέπει από την Γαλλία να του έχουν χορηγήσει τον αριθμό κοινωνικής ασφάλισης κλπ. Έχουν πολύ περιορισμένοι λοιπόν. Επίσης ε, ζήτημα έχουμε και με το Smart Grid για την βελτίωση της ε, περιβαλλοντικής, ε, του περιβαλλοντικού σχεδιασμού για τα κτίρια. Η NEA ουρανή, single sky, οι ποτάμιες μεταφορές, τα ηλεκτρονικά μητρώα για τους για τους χρήστες των οδικών μεταφορών ή των οδικών κόμβων καλύτερα, των οδικών, του οδικού δικτύου και επίσης σημαντικό ρόλο παίζει σε όλα αυτά η επικοινωνία, η ανταλλαγή των πληροφοριών. Το πιο σημαντικό ίσως να είναι η έννοια της ασφάλειας στην κοινωνία της πληροφορικής. Χρειάζεται η προστασία των κρίσιμων υποδομών, της τεχνολογίας των πληροφοριών, των, τηλεπικοινωνιών που αποτελούν μέρος της κρίσιμης τεχνολογίας, ε, υποδομής, έτσι ώστε να προστατεύουμε και τον καταναλωτή για να έχουμε, και αυτό σημαίνει να έχουμε και ακαιρεότητα και διαθεσιμότητα και αυθεντικότητα, έλεγχο ε, ε γνησιότητα των στοιχείων. Ίσως μπορούν να μας πούν οι συνάδελφοι μερικά πράγματα λίγο για την ε, αμοιβαία αναγνώριση ηλεκτρονικής υπογραφής τι έχει γίνει. Ο Πρόεδρος. Κύριε Καβάλιο, ευχαριστώ. Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω την Πιλάρ Δελ Καστίγιο για την πολύ καλή δουλειά που έκανε και να τονίσω το εξή: Το θέμα των αρμοδιοτήτων. Θεωρώ ότι υπάρχουν δύο επίπεδα αρμοδιοτήτων. Υπάρχει η γενική αρμοδιότητα. Sorry. And you have the very high skilled... του γενικού πληθυσμού, του γενικού κοινού. Αν θέλετε και υπάρχουν και ε, οι συγκεκριμένες ικανότητες των ε, ειδικών, των ε, μηχανικών. Αυτό μας λείπει στην Ευρώπη. Χρειαζόμαστε πιο πολλούς μηχανικούς. Ε, έχουμε πολλούς ε, νέους που δεν έχουν δουλειά, αλλά όχι στον τομέα αυτό. Θα πρέπει λοιπόν να προσελκύσουμε πιο πολλούς ε, φοιτητές στον τομέα της μηχανικής των υπολογιστών και ο λόγος που έχουμε τέτοιο έλλειμμα είναι διτός. Καταρχάς η χαμηλή απόδοση που υπάρχει γενικά στη φυσική και στα μαθηματικά. Θα πρέπει λοιπόν να προωθήσουμε τα μαθηματικά τη φυσική στις νεαρές ηλικίε, προκειμένου να τα επιλέξουν τα παιδιά αυτά και σε μετέπειτα φάσεις. Και ο δεύτερος λόγος είναι ότι προς το παρόν οι πιο πολλές τα πανεπιστήμια είναι οι γυναίκε. Ο μεγαλύτερο αριθμό είναι οι γυναίκες. Και οι γυναίκε σπάνια επιλέγουν τι ε, κατευθύνσει αυτέ. Άρα η αναλογία ανδρών και γυναικών σε τέτοιε επιστήμες ε, μηχανική υπολογιστών είναι 5 προς 1. Επίσης, θα πρέπει να προσελκύουμε τα άτομα υψηλή εξειδίκευση από όλο τον κόσμο, Όπω γίνεται στην Καλιφόρνια για παράδειγμα, αλλά αυτό θα αποτελέσει μεγάλη δυσκολία για πολλά κράτη-μέλη. Γιατί υπάρχει μια ολόκληρη γραφειοκρατία η οποία δεν είναι εύκολο να ξεπεραστεί. Άρα ο κόσμος τελικά καταλήγει πιο εύκολα στις Ηνωμένε Πολιτείε παρά στην Ευρώπη. Επίσης, όπως αναφέρθηκε ήδη, θα πρέπει να υπάρχει να υπάρχουν άτομα καλά, καλ, υψηλής εκπαίδευσης. Θα πρέπει λοιπόν να προωθήσουμε την έρευνα και κυρίως τον σύνδεσμο μεταξύ ε, έρευνας επιχειρήσεων και καινοτομία. Θα ήθελα λοιπόν αυτά να τονιστούν λίγο πιο έντονα στην έκθεση. Ευχαριστώ. Κύριος Βέιμπερ, λέει ο Πρόεδρος. Εγώ θα έλεγα εισαγωγικά ότι το θέμα που με εξαιρετικό τρόπο εξέτασε η συγγήτρια είναι ένα από τα πιο σημαντικά θέματα της σημερινής εποχής. Πρόκειται για μία επανάσταση, ψηφιακή επανάσταση που θα έχει τις ίδιες επιπτώσεις με την εφεύρεση της τυπογραφίας κάποτε. Ο τρόπος κατανάλωσης εργασίας, επικοινωνίας και σκέψης επηρεάζονται. Εμείς βρισκόμαστε στην αρχή αυτής της ψηφιακής επανάστασης και προχωράει πάρα πολύ γρήγορα και η ικανότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μείνει στην αιχμή αυτού του κινήματος ε, είναι σημαντικότατη για το μέλλον της Ένωσης. Από δύο φόρο τιμή στην έκθεσή σας και στην ευρύτητα του πνεύματός σας, διότι πραγματικά το, βάζετε το, τη θεματική αυτή στο πραγματικό της ύψος όπως είπε και ο κύριος Λαμπέρ, είμαστε ήδη καθυστερημένοι. Το χάσμα μεγαλώνει μεταξύ ημών της Ιαπωνίας και των Ηνωμένων Πολιτειών. Και όχι απρός, εμείς πρέπει να βρισκόμαστε στην αιχμή αυτών των τεχνολογικών ορίων που ε, ορίζονται αλλά να ξεπεράσουμε και το χάσμα που μεγαλώνει. Η βάση λοιπόν της εκθεσής σας είναι εξαιρετική. Δύο σημεία γιατί δεν έχουμε χρόνο να μπούμε σε λεπτομέρειες. Θα ήθελα διευκρινήσεις για το άρθρο 19, δηλαδή στο να προχωρήσει πιο γρήγορα η συζήτηση για τα πνευματικά δικαιώματα στην Ευρώπη, κατά πολέμηση της πειρατείας, είναι πολύ σημαντικό αυτό, μας τυχιώνει εδώ και χρόνια και στο 118 άρθρο της ε, λειτουργίας ε, της ε, Ένωσης το άρθρο αυτό θεωρώ ότι έχει ξεπεραστεί δηλαδή να έχουμε πνευματικά δικαιώματα στη βάση της επικουρικότητας χρειάζονται ευρωπαϊκά δικαιώματα και ε, περιπτώσει εγώ διαφωνώ σε αυτό το άρθρο 19 και στα ευρωπαϊκά πνευματικά δικαιώματα. Χρειάζεται λοιπόν και αυτό να το αναπτύξουμε. Εμείς ε, θα πρέπει να έχουμε κατά νου τις νέες γενιές οι οποίες έχουν μια φυσιολογική τάση προς αυτές τις νέες τεχνολογίες ε, και όχι απλώς εμείς να, να, να απαιτήσουμε δηλαδή να έχουν αυτές τις τεχνολογίες τα σχολεία αλλά δείτε τι γίνεται ας πούμε στις σκανδιναβικές χώρες όπου με, που τα, με το που τα παιδιά μπαίνουν στο γυμνάσιο τους δίνουν έναν υπολογιστή ενώ παλιά τους δίναν τα βιβλία Πρέπει λοιπόν εμείς να εκμεταλλευτούμε αυτό το φθόρμητο κίνημα το νέο της νέας γενιάς. ευχαριστώ. Θα ήθελα να κάνω δύο σχόλια σύντομα. Καταρχάς να υποστηρίξω κάτι που είπε ο συνάδελφος, η συνάδελφος κυρία Βαλεάν. Είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι χρειαζόμαστε ρύθμιση προκειμένου να προωθήσουμε τον ανταγωνισμό. Καταλαβαίνουμε φυσικά ποιο είναι ο στόχος μας. Θέλουμε να υπάρχει πλήρη ανταγωνιστικότητα στην αγορά τηλεπικοινωνιών. Γιατί αυτό ωφελεί και τις επιχειρήσεις και τους πολίτες. Έχουν ε, όσο το δυνατόν πιο πολλές ε, επιλογές γίνεται και στις καλύτερες δυνατές τιμές. Χρειαζόμαστε όμως το ρύθμιση για να το πετύχουμε αυτό. Και γιατί χωρίς ε, ρύθμιση οι φορεί θα καταλήξουν σε καθεστώ κυριαρχίες αν θέλετε στην αγορά το οποίο δεν θα είναι δίκαιο. Και αυτό θέλουμε να το αποφύγουμε. Κατά δεύτερον, να συμφωνήσω με την εισηγήτρια ότι δεν θέλουμε να ξανανοίξουμε το πακέτο για τις τηλεπικοινωνίες. Τώρα θα πρέπει να εστιαστούμε, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, ε, στην ε, πλήρη εφαρμογή του πακέτου αυτού και μάλιστα σε διεθνές επίπεδο. Και αυτό περιλαμβάνει και τον λειτουργικό διαχωρισμό που έχει αποδεχτεί σε πολλά κράτη-μέλη ότι είναι πάρα πολύ αποδοτικό σε ό,τι αφορά την ε, εγκαθίδρυση καθεστώτο ανταγωνισμού. Άρα, συμφωνώ να μην ξανανοίξουμε το πακέτο αυτό, να κινηθούμε προς τα εμπρός. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Τώρα, συνάδελφοι, ακούσαμε την άποψη του Κοινοβουλίου. Να δώσουμε τώρα τον λόγο στον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Η συζήτηση φτάνει σε μια πολύ χρήσιμη για μας στιγμή και θα βοηθήσει πολύ, θα εμπλουτίσει κατά αυτόν τον τρόπο τις συζητήσεις εσωτερικές στην Επιτροπή. Όπως ξέρετε η Επιτροπή θα προσδιορίσει τις θέσεις, τις προτάσεις της, την προσέγγιση της στην ψηφιακή ατζέντα, αλλά έχει ταυτόχρονα επισημάνει ξεκαθαρό ότι δεν πρόκειται να το πράξει αυτό πριν ακούσει και την έποψη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Το χρονοδιάγραμμα στο το οποίο έχουμε προσδορίσει αυτή τη στιγμή είναι ότι θα υιοθετήσουμε την έκθεση το Μάρτιο. Τον Απρίλιο θα έχουμε σημαντική ε, συνεδρίαση που οργανώνει η Ισπανική Προεδρία όπου θα συζητήσουν το ίδιο θέμα λίγο πολύ οι Υπουργοί και κυκλοφορεί και ένα έγγραφο για την στρατηγική και μόνο αφού θα έχουμε λάβει ε, τις ε, παρεμβάσεις αυτές θα καταλήξει η Επιτροπή. Αυτή είναι η κατάσταση λοιπόν και θα ήθελα να υπογραμμίσω ε, Επιτρέψτε μου να διατυπώσω κάποιες προσωπικές παρατηρήσεις για, τις, ε, για την έκθεση κυρίας Δικαστήριο. Θα ήθελα να υπογραμμίσω τις ε, δύο μεγάλες προκλήσεις που είχε να αντιμετωπίσει και που σημαίνουν για το έγγραφο το δικό μας ε, γιατί το σημαντώσουμε και αυτό ότι αποστέλλεται ένα μήνυμα στην κοινή γνώμη αλλά και στους, στους πολιτικούς ότι χρειάζεται κάτι να γίνει, χρειάζεται να επενδύσουμε πολύ περισσότερο στις ε, ψηφιακές τεχνολογίες να αποκομίσουμε το μέγιστο δυνατό από τις τεχνολογίες αυτές τώρα και γιατί τώρα και όχι πριν από μερικά χρόνια, γιατί τις τεχνολογίες αυτές είχαμε εδώ και καιρό στη θέση μας. Ο κύριος Λάμπρεχτς επεσήμανε κάποιους από τους κύριους λόγους για τον οποίους τώρα πρέπει να καταβάλουμε μια ιδιαίτερη προσπάθεια. Υπάρχει όμως μια πρώτη ε, πρόκληση που την έχουμε αντιμετωπίσει και η άλλη πρόκληση είναι πώς καταγράφουμε, εξηγούμε καταστάσεις όπου αντικειμενικά πρέπει να παρεμβαίνουμε σε πολλούς πολλούς τομείς. Πολύ περισσότεροι τομείς πώς θα μπορούσαν να ε, απαριθμιστούν σε μια πολιτική ε, συζήτηση. Δηλαδή πλέον πρέπει σε 50, 60, 70 επιμέρους παιδεία να αναλάβουμε δράση. Αλλά βέβαια σε μια πολιτική συζήτηση πρέπει να είμαστε θέσει να διατυπώσουμε ταχαίως ένα ε, πολιτικό μήνυμα και αυτό δεν, μπορεί να γίνει αν αναφερθούμε σε 60-70 διαφορετικά πεδία. Η κυρία Ντεκαστήγιο έχει κάνει μια πολύ καλή δουλειά πιστεύω. Έχει βοηθήσει πολύ αν και κάποιες άλλες ε, κάποιες παρεμβάσεις ε, ζητούν ζητούν να επεκταθεί και σε άλλα θέματα. Δεν πρέπει να λησμονούμε όμως ότι και η πρόταση της Μαδρίτης έγινε δεκτή τον Ιανουάριο από το χώρο, τον οικονομικό, από τις επιχειρήσεις που είπαν τι θα πρέπει να είναι η ε, ηλεκτρονική ατζέντα με 78 συστάσεις. Πράγμα που δείχνει πόσο ε, περίπλοκο είναι το ζήτημα. Και ναι, βεβαίω, όταν μιλούμε για τεχνολογίε πληροφορία και τηλεπικοινωνία, πρέπει να υπάρχει τη επικοινωνία μα. Πρέπει να υπάρχει δηλαδή το δίκτυο. Και άπαξ και υπάρχει το δίκτυο, αναπτύσσουμε τι δυνατότητε και τα διάφορα ζητήματα τα οποία πρέπει να καλυφθούν φερρυπίν ικανότητα χρήση των τεχνολογιών, εμπιστοσύνη, δηλαδή αίσθηση ασφάλειας, προστασία προσωπικών δεδομένων κτλ. Και πολλοί άλλοι τομείς που ακολουθούν, εσωτερική αγορά, δηλαδή η πληροφορία, η, τεχνολογία της πληροφορίας και των τηλεπικοινωνιών μας δείχνει και ποιες είναι οι ελλείψεις μας ε, στην κοινή αγορά. Μειώνονται οι αποστάσεις ε, ε, πέφτουν οι φραγμοί ή τα όρια χάρη στην τεχνολογία της πληροφορίας των τηλεπικοινωνιών και βλέπουμε τι ε, κενά έχουμε και που πρέπει να κάνουμε πιστή προσπάθεια και για την επιστήμη και για την έρευνα και για την αποτελεσματικότητα της ενέργειας και για την βιώσιμη ανάπτυξη. Αυτή είναι πολλοί οι τομείς στους οποίους μπορούμε να αξιοποιήσουμε αυτή τη νέα τεχνολογία ε, προς όφελός μας. Δεν θα υπησέλθω στις διάφορες ε, λεπτομέρειες της έκθεσης, ασφαλώς μας στη σε κάθε σχόλιο. Ε, ήθελα να υπογραμμίσω μια παρατήρηση που διατύπωσαν αρκετοί βουλευτε ότι η έκθεση δεν θα πρέπει να θεωρηθεί ως ευκαιρία για αναθεώρηση του ε, ρυθμιστικού πλαισίου. Δεν μπορεί δηλαδή η ψηφιακή ατζέντα να αποτελέσει λόγο α, ανατροπής του ρυθμιστικού ψηφίου. Αυτό, πλαισίου. Αυτό είναι βέβαια αυτονόητο κατά με αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει και να υπογραμμίσουμε το δεδομένο αυτό, γιατί βρισκόμαστε σε μία κατάσταση όπου η εξέλιξη των δικτύων είναι πολύ βραδύτερη από ό,τι θα θέλαμε. Και ο κύριος λόγος είναι η ε, απόδοση των επενδύσεων, οι επενδύσει που κάνουν επιχειρήσει και αποδόση που μπορούμε να αναμένουμε από τι επενδύσει αυτέ. Και πολλά μπορούν ακόμη να πράξουν τα κράτη-μέλη ώστε να μειώσουν αυτό το, ε, αυτές τις επενδύσεις. Το μήνυμα λοιπόν που θα πρέπει όλοι μαζί να αποστείλουμε είναι ότι έχει προσαρμοστεί το ρυθμιστικό πλαίσιο, έχει διασαφινιστεί, υφίσταται, λειτουργεί. Κλείνει αυτή η συζήτηση. Αυτό θα είναι το ρυθμιστικό μας πλαίσιο για τα επόμενα χρόνια και πολλά ακόμα μένει να, μένουν να γίνουν από τα κράτη-μέλη για να μειωθεί το κόστος των επενδύσεων. Φερρυπίν. Ε, δικαιώματα πρόσβασης, υποδομής, προσαρμογή των διαφορών κωδικών, κωδίκων μάλλον. Ε, όλα αυτά τα θέματα στα οποία θα πρέπει να δώσουμε την έμφαση για, τις, για τα επόμενα χρόνια. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Σάντι και μετά η συγκεκριά, παρακαλώ. Se trata de reiniciar eh, de nuevo un debate. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Για να κλείσουμε μόνο, δεν θέλω να ξανανοίξω μια συζήτηση που έχει γίνει εδώ και πολλέ φορέ. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσε όλε τι παρεμβάσει και ευχαριστώ ιδιαίτερω ε, και του ε, εισηγητέ, τον εκπρόσωπο της, και του εισηγητέ και τον κύριο Κολασάντε από την Επιτροπή. Για να κλείσουμε λοιπόν το θέμα, θα ήθελα να πω δύο-τρία πράγματα. Καταρχά, ότι είμαστε, πιστεύω, σε κοινή πιστεύω γραμμή πράγμα το οποίο με χαροποιεί ιδιαίτερα και από αυτή την έννοια δεν με εκπλήσει η διαπίστωση αυτή, διότι είναι πολύ ο καιρό που συζητούμε ακριβώς τα θέματα της αναθεώρησης νομοθεσίας του τομέα αυτού, δύο χρόνια και παραπάνω ίσως. Μας απασχολεί το θέμα αυτό και η Επιτροπή μας λίγο πολύ αρχίζει να δημιουργεί μέσα στους, στους κόλπους της Επιτροπής να δημιουργείται ένα κοινό ακαδημαϊκό θα έλεγα πλαίσιο, μια, ένα κοινό δόγμα, μια κοινή θεωρία και με τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μπορούμε να έχουμε μια ε, συνεκτική στάση. Πολλά είναι τα θέματα, οι τοποθετήσεις στις οποίες ε, συμμερίζονται όλες οι πολιτικές ομάδες, πράγμα το οποίο είναι πολύ σημαντικό, για να αρχίσουμε να πραγματοποιούμε τα προσεχή βήματα την ώρα του προσδιορισμού της ψηφιακής ατζέντας. Και θα ήθελα να ε, επιμείνω ιδιαίτερω ε, στα τελευταία λόγια του κ. Κολασάντη, τα δικά μου επίση τελευταία λόγια, αλλά και κάποιων άλλων συναδέλφων που έλεγαν το λόγο εδώ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και εν γέννη νομίζω ε, δεν ε, έχει τύχει ενδεχομένως κάποτε κάπου να υπόθηκε μια κουβέντα αλλά ε, ποτέ δεν αμφισβητήθηκε το, αμφισβητήθηκε το πεδίο αυτής της έκθεσης ή δεν έγινε μια προσπάθεια να αναμειχθεί με κάποια άλλα ε, παιδεία, όπως είπε ο κ. Κροσάντη νωρίτερα, το τομέα των τηλεπικοινωνιών κτλ. Και επίσης, δεν θέλω να σημειώσω ότι για κάποιες από τις παρεμβάσεις, τον κύριο Λάμπερτ παραδείγματος χάρη, ήταν πολύ χρήσιμη, πολύ ενδιαφέρουσα η παρέμβασή σας και δεν μπορώ να συμφωνήσω περισσότερο. Και δεν μπορώ να συμφωνήσω περισσότερο, όχι μόνο θεωρητικά, αλλά στα όσα πράγματι λέγεται, γιατί αυτά είναι ακριβώ και τα επιχειρήματά μου, ότι θα πρέπει να έχουμε μια προσέγγιση ε, για τις τηλεπικοινωνίες ε, και την ε, πληροφορία Και εγώ αναφέρομαι παραδείγματι στο ICT Policy Stream, τη δυνατότητα δηλαδή που μπορούμε να έχουμε ε, στην κοινωνία της πληροφορίας να διατρέξουμε ολόκληρη την βιομηχανία, να επιτρέψουμε δηλαδή σε όλο το χώρο τον οικονομικό, τον επιχειρηματικό, να αξιοποιήσει αυτές τις δυνατότητες. Και εδώ μιλώ για διάφορους τομείς επιχειρηματικής δράσης, οικονομικής δράσης, συμπεριλαμβανομένων και των, ε, συμπεριλαμβανομένης και της ενέργειας, γιατί μπορούμε να συνδυάσουμε την ICT με την ενέργεια χαμηλής ε, χρήσης άνθρακα. Πρέπει να δούμε λοιπόν ποιοι είναι οι συσχετισμοί και πώς, ε, μπορεί να συμπράξουν, πώς μπορούν να συμπράξουν διάφοροι κλάδοι του επαγγελματικού ή βιομηχανικού χώρου, παραγωγικού χώρου. Ποια θα είναι η αναλογία παρέμβασης της ε, διοίκησης, ε, το switch-over το, της ε, διοίκησης στην ψηφιακή εποχή, ο χάρτης των δικαιωμάτων των χριστών, εγώ ζητώ να θεωρώ ότι υπάρχει ανάγκη και ένα χάρτη δικαιωμάτων των χριστών, όλα αυτά λοιπόν τα ζητήματα τα οποία συμμερίζομαι και εγώ και 100% συμφωνώ, μπορώ να το πω απερίφραστα στο σημείο αυτό. Φυσικά η σαφή συγκεκριμένη διατύπωση που χρησιμοποιείται πάντοτε ε, χρήση βελτιώσεως ή χωρί βελτίωση στην ισχύουσα διατύπωση και γι' αυτό ευχαριστώ πολύ για την παρέμβασή σας και για τις παρατηρήσεις σας. Εδώ έχουμε να κάνουμε μια πρώτη σκέψη και ιδέες που διατυπώνουμε με την έκθεση και για το ζήτημα του ευρωπαϊκού copyright, τη της προστασίας των ευρωπαϊκών δικαιωμάτων πραγματικής ιδιοκτησίας. Ναι, ίσως πρέπει να είμαι κοντά στο μικρόφωνο για να μιλάω. Είναι ένα πολύ περίπλοκο θέμα είναι πολλές ιδιαιτερότητες στους τομείς που θα μπορούσαν να υπαχθούν στην έννοια της προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων, πνευματική δημιουργία, οπτικοακουστικά μέσα κτλ. Πιστεύω ωστόσο, χωρίς να έχω όμως απόλυτες θέσεις, πιστεύω ότι είναι ένα ζήτημα το οποίο θα έπρεπε να παραδεχθούμε ότι αξίζει να συζητηθεί. Είναι περίπλοκο. Αν όμως θέλουμε να μιλάμε για μια ενιαία ψηφιακή αγορά, δεν μπορεί να παραμείνει το θέμα αυτό στο περιθώριο. Ή να το εξετάσουμε μόνο ακροθυγός. Άλλωστε αυτό έχω ήδη συμπεριλάβει και στην έκθεση ε, με αυτό το νόημα. Βεβαίως ίσως χρειάζονται περισσότερες ε, νέε ιδέες ως προ τη διατύπωση τη συγκεκριμένη συγκεκριμένης ε, στόχευση. Κατά τα άλλα, ευχαριστώ πάρα πολύ τους πάντες για την συζήτηση. Με βοήθησε πολύ, μου έδωσε πολλές νέες ιδέες και βέβαια το επόμενο στάδιο θα είναι τροπολογία. τροπολογίες. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Κλείνουμε λοιπόν και αυτό το σημείο στην ημερήσια διάταξη. 11 Φεβρουαρίου, 12 η ώρα το μεσημέρι, είναι η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών. Και τώρα παρακαλέσω να παρακαλέσω να περάσουμε στο επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη. Λυπάμαι, συνάδελφοι, που έχετε μόνο 15 λεπτά στη διάθεσή σας. Νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το επιλύσουμε επί της αρχής. Πώς μπορούμε να λύσουμε αυτό το θέμα προκειμένου όλες οι εκθέσεις να έχουν το ίδιο χρόνο στη διάθεσή τους, να μην ρίχνονται οι τελευταίες εκθέσεις. Μιλάμε για την έκθεση αυτή. Θα πρέπει να συζητηθεί σε 15 λεπτά. Να δώσω το λόγο στον εισηγητή. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα κάνουμε μια προσπάθεια να βγάλουμε πέρα. Εν συντομία. η σχέδια, το σχέδιο οδηγία για τις καθυστερήσεις πληρωμών στις εμπορικέ συναλλαγές υποβλήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Απρίλιο του 2009 και η πρόταση περιλαμβάνεται σε ένα ευρύτερο πακέτο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αυτό το Small Business Act όπως το λέμε. Προτού περάσω σε στοιχεία ε, επί του περιεχομένου, θα πρέπει να πω ότι πρόκειται για μια νέα έκδοση του κειμένου της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Υπάρχει μια παλιά οδηγία η οποία δυστυχώς δεν πέτυχε τους ε, στόχους ε, που είχαν τεθεί. Θα βασιστώ στα στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας. Το Δεκέμβριο Κοίταξα τα στοιχεία αυτά, τα οποία αφορούν συγκεκριμένα προβλήματα στην Ευρώπη. Πρόκειται για ένα πρόβλημα που επηρεάζει ιδιαίτερα πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις μικρές επιχειρήσει. Α, συγγνώμη, λέει ο Πρόεδρος μήπως ε, θα μπορούσαν να βγουν έξω όσοι ενοχλούν, παρακαλώ, τον εισηγητή. Να μην γίνονται συζητήσει και πηγαδάκια μέσα στην αίθουσα. Ευχαριστώ. Ωραία. Ιδιαίτερα λοιπόν στην φάση της κρίσης που διανύουμε θα μπορούσε να έχει ιδιαίτερα αρνητικό αντίκτυπο αυτό σε ό,τι αφορά πολλές μικρές επιχειρήσεις που κινδυνεύουν να κλείσουν, να πτωχεύσουν. Και αυτό φυσικά συνεπάγεται προβλήματα με τη σειρά του για την απασχόληση. Κανείς λοιπόν δεν μπορεί να παραγνωρίσει ε, τη σημασία της νομοθεσίας αυτής. Υπάρχει ανάγκη να ληφθεί γρήγορα και αποτελεσματικά δράση για να δοθούν απαντήσεις στα προβλήματα τα οποία ταλανίζουν τις επιχειρήσεις αυτές στη δύσκολη αυτή η οικονομική περίοδο. Η πρόταση λοιπόν της Ευρωπαϊκής Επιτροπής συνοψίζεται σε τέσσερα σημεία. Καταρχάς, σε ό,τι αφορά τις ε, συναλλαγές μεταξύ των ιδιωτικών σημαντικών ε, φορέων και σε ό,τι αφορά το χρόνο πληρωμών και την έλλειψη οποιαδήποτε σημαντικού ορισμού για, τη σημαντική, για την πληρωμή αυτή. 30 ημέρες ισχύουν ως όριο. Κατά δεύτερον, οι συναλλαγές με τη δημόσια δίκηση. Και πάλι 30 ημέρες είναι η προθεσμία μετά την παραλαβή του τιμολογίου. Ωστόσο, η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και νομίζω ότι αυτό αποτελεί και το όριο, ε, δίνει πολλές ε, περιπτώσεις εξαιρέσεων. Και αυτό ασφαλώς συνεπάγεται ένα 5% επιπλέον σε σχέση με το επιτόκιο που υποβάλλεται. Υπάρχουν κάποιες ρήτρε προφανώς ε, σε συμβάσεις. Το τέταρτο σημείο τώρα, το οποίο αποτελεί τον ορισμό των αποζημιώσεων σε περίπτωση καθυστέρησης πληρωμών Τα άρθρα αυτά προφανώς επηρεάζουν την ε, διαφάνεια, όπως και στην προηγούμενη οδηγία και αφορούν κυρίως ε, τους ορισμούς προς την κατεύθυνση αυτή. Άρα, βάσει της συζήτησης που έγινε στην Επιτροπή το Δεκέμβριο και εν ώψη των δικών μου απόψεων και των σκιωδών. Η συζήτηση θα πρέπει να γίνει κυρίως ε, με τους ε, συναδέλφους για τα θέματα πιο, τα, τα, τα, πιο ανοιχτά. Λοιπόν, εγώ είχα συναντήσεις με την εισηγήτρια την κυρία Βάιλερ και εξέτασα ε, την εργασία της αλλά άκουσα και τις ακροάσεις ε, ε, στην Επιτροπή μας κυρίως η ακρόαση εκείνη με τους εκπροσώπους των Εθνικών Κοινοβουλίων γιατί αυτή η οδηγία βαραίνει διαφορετικά στα 27 κράτη της Ένωσης. Εγώ πιστεύω ότι δεν υπάρχουν προβλήματα και γιατί το πόσο είναι πήγους αυτή η πρόταση οδηγίας. Αυτό το κείμενο έτσι όπως έχει κατατεθεί στο Κοινοβούλιο. Είναι ένα κείμενο το οποίο μπορούμε να συμμεριστούμε. Θεωρώ μόνο ότι χρειάζονται μενικές μικροαλλαγές για να υπάρχει μια νομική ασφάλεια σε αυτή την οδηγία και για να αποφύγουμε τον κίνδυνο να ξαναπέσουμε σε αυτές τις ε, δυναμικές, ε, ερμηνευτικές δυναμικές ε, και στις παρεκκλήσεις που είχαμε στην 35 του 2000 Γι' αυτό, γι αυτό φτάνουμε δηλαδή και στην επανεξέταση αυτής της οδηγίας. Λοιπόν, πρώτο, συναλλαγές μεταξύ των επιχειρήσεων, business to business. Είναι πολύ αδύναμη πρόταση οδηγίας για αυτό το σημείο. Γιατί είναι οι ιδιώτες που έχουν την εντολή για την καταβολή των πληρωμών. Και αυτό βαραίνει αρνητικά ε, τις διαπραγματευτικές δυνατότητες των ιδιωτών και οι πιο μικρές επιχειρήσεις ε, μπορούν ε, να δεχθούν συμβα... συμβάσεις οι οποίες να είναι ιδιαίτερα επιβαρυντικές για αυτές. 60, χρόν... 60 μέρες λοιπόν πληρωμές για τους ιδιώτες. Τώρα για 30 μέρες για τους δημοσίους οργανισμούς και να περιορίσουμε δραστικά την παρέκκληση. Μόνο μία παρέκκληση δικαιολογημένη ανάλογα με την αναγκαιότητα χωρίς όμως ποτέ υπέρβαση των 60 ημερών. Μία λύση επίσης που να συμπεριλαμβάνει και τις ε, ε, επιχειρήσεις κοινή ωφελίας. Ε, επίσης, αποζημίωση για τις δαπάνες. Η αποζημίωση δηλαδή των προσφυγών που κάνει κανείς για να ξαναπάρει πίσω τα λεφτά του πρέπει να είναι εκτελεστικές για να αποφεύγουμε στρεβλώσεις. Επίσης, τελευταίο, η πληροφόρηση. Εγώ πιστεύω ότι είναι ένα σημείο πάρα πολύ σημαντικό, διότι δεν μπορεί να υπάρξει καταπολέμηση των καθυστερημένων πληρωμών χωρίς να υπάρχει πληροφόρηση, δηλαδή να αποκτήσουν συνέστηση και οι επιχειρήσεις για τα νέα τους δικαιώματα. Εγώ πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό και για αυτή την Επιτροπή να παρακολουθήσουμε από κοντά τη σωστή διάδοση της πληροφόρησης μεταξύ επιχειρήσεων και κοινωνίας ενημερώνοντας όλους για τα πλεονεκτήματα αυτής της οδηγίας. Εγώ, Πρόεδρε, με πρόθεση δεν εξέτασα ένα ειδικό θέμα της οδηγίας. Είναι πολύ σημαντικό και το θεωρώ ιδιαίτερα ε, ευαίσθητο λόγω της επιρροής που μπορεί να έχει στον προϋπολογισμό, στους εθνικούς προϋπολογισμούς. Στην παράγραφο 5 του άρθρου 5 όπου έχουμε όπου όταν έχουμε ε, χρέη και απέτηση χρεών εμείς ε, ζητείτε μάλλον αποζημίωση ε, από τον δημόσιο οργανισμό ή τις δημόσιες υπηρεσίες αντίστοιχη του 5% του αρχικού ποσού του χρέους. Εγώ το σκέφτηκα πολύ αυτό και πιστεύω ότι πρέπει να ξαναεξετάσουμε αυτή την παράμετρο. Αυτή η οροφή του 5% είναι πολύ ψηλή. Χρειάζεται λοιπόν να ξαναδούμε αυτή την οροφή, να την μειώσουμε και να επεκταθεί και στις συναλλαγές μεταξύ ιδιωτών, ούτως ώστε οι καθυστερήσεις των πληρωμών να μην ε, εμπίπτουν μόνο στο δημόσιο τομέα. Λοιπόν, εγώ περιμένω τις απόψεις σας και ελπίζω να βρούμε μια σωστή λύση που θα λαμβάνει υπόψη όσα θα πούνε οι συνάδελφοι. Θέλω να ευχαριστήσω τους και ηγητές για τη δουλειά τους μέχρι τώρα και παρακαλώ σε μια επόμενη συνεδρίαση μεταξύ ημών και άτυπη ε, τον ορισμό ορισμένων συμβιβαστικών τροπολογιών που είναι απαραίτητες για την ολοκλήρωση των εργασιών μας. Thank um, Σας ευχαριστώ. Εγώ μιλώ εξ ονόματος του κυρίου Ρόντε, ο οποίος είναι ο σκιώδης εισηγητής για το θέμα αυτό. Εν γέννη υποστηρίζουμε τις θέσεις και το σχέδιο του εισηγητή. Είναι καλά ισορροπημένο το κείμενο και περιλαμβάνει σωστές ε, διευκρινήσεις και ενισχύει κάποιες βασικές ε, διατάξεις. Σωστό. Συμφωνούμε γενικά με τις τροπολογίες του εισηγητή για να ενισχυθούν οι διατάξει που αφορούν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε ό,τι αφορά το εμπόριο μεταξύ των επιχειρήσεων, γιατί πολλές φορές βλέπουμε κατάχρηση της κυριαρχούσα θέση των μεγάλων επιχειρήσεων, μονομερό. Ωστόσο, συνειδητοποιούμε και αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχει ανάγκη να διατηρήσουμε και το συμβατικό δικαίωμα των επιχειρήσεων. Πιστεύουμε ότι θα πρέπει να βρεθούν λύσεις προκειμένου να ανταποκριθούμε σε αυτές τις ελαφρώς αντικρουόμενες ε, θέσεις. Μιλήσατε για τις μεγάλες επιχειρήσεις που θα πρέπει να μην έχουν τη δυνατότητα αναδρομικά να αλλάζουν τις, ε, τους όρους πληρωμής μονομερός. Ίσως λοιπόν θα πρέπει να συμπεριληφθούν διατάξεις στην οδηγία που θα δώσουν αντικίνητρα σε ό,τι αφορά μονομερείς ε, και αναδρομικές αλλαγές των όρων πληρωμής. Τέλος, να αναφέρουμε ότι συμφωνούμε με την ενίσχυση των διατάξεων σε ό,τι αφορά τις ε, προμήθειες προς την κυβέρνηση, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την μείωση του εύρους των εξαιρέσεων. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Επόμενος ομιλητής, ο κ. Μπένσον. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω για την καλή δουλειά που έχει γίνει στο σημείο αυτό. Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό θέμα, άλλωστε. Τη Δευτέρα έγινε μια τέτοια συζήτηση και όλοι είπαν ότι πραγματικά πρόκειται για ένα μεγάλο πρόβλημα που είναι ιδιαίτερα σημαντικό στην παρούσα κρίση. Το γεγονός δηλαδή ότι υπάρχουν μεγάλες καθυστερήσεις στις πληρωμές. Και θα ήθελα να υπογραμμίσω το εξής. Μεταξύ των ε, δημόσιων και ιδιωτικών φορέων υπάρχουν μεγάλες, πληρω... μεγάλες καθυστερήσεις και μεγάλα προβλήματα στις πληρωμές και μεγάλες επιχειρήσεις υποχρεώνονται να αποδέχονται όρους συμβατικούς ε, ε, μειονεκτικούς λόγω της κρίσης. Οι μικροί λοιπόν ε, καταπιέζονται από τους μεγάλους και σε αυτές τις εποχές όπου οι τράπεζες επιβάλλουν αυστηρά μέτρα, ο αντίκτυπος πλήττει τελικά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δεν έχουν άλλο τρόπο να αμυνθούν. μεταξύ των ιδιωτικών εταιριών υπάρχουν συγκεκριμένοι όροι για τις συναλλαγές, οι οποίοι όμως δεν ισχύουν μεταξύ δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Ίσως λοιπόν θα έπρεπε να οριστεί και αυτός ο κλάδος για τις σχέσεις μεταξύ ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. Θεωρώ ότι πραγματικά είναι σημαντικό να εφαρμοστεί σωστά η οδηγία αυτή γιατί κοιτώντα την προηγούμενη οδηγία διαπιστώνουμε ότι πολύ απλά δεν λειτουργήσε και βρισκόμαστε σε μια κατάσταση όπου οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ευρωπαϊκής οικονομίας υπόκεινται τέτοια πίεση από τις μεγάλους ε, φορείς που τελικά κινδυνεύουν. Χαίρομαι λοιπόν που θα γίνει η συζήτηση αυτή προκειμένου να ανταλλάξουμε απόψεις. Οι διατάξεις αυτές πραγματικά θα πρέπει να αποβούν προ όφελο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Είναι ένα τεράστιο πρόβλημα το οποίο δεν θα λυθεί από μόνο του, θα διαγωθεί περαιτέρω. Η όλη συζήτηση αναφορικά με τις δημόσιες προμήθειες, τις ιδιωτικές προμήθειες. Όλα αυτά ε, είναι στοιχεία που έχουν ρόλο, έχουν ε, σημασία για τη συζήτηση και οι πτυχές αυτές καταδεικνύουν μάλλον μας ε, οδηγούν στη σωστή κατεύθυνση. Δεν θα πρέπει να υπάρχει διαφορά μεταξύ δημοσίου κλάδου και μεγάλων ιδιωτικών επιχειρήσεων. Και χαίρομαι που έχει ξεκινήσει αυτή η συζήτηση. Ευχαριστώ, κύριε Μπιουτικόφερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να απαντήσω απευθείας, να συνεχίσω μόνο απευθείας τόσο είπε ο προλαλή διότι πιστεύω ότι θα πρέπει και εμείς να μεριμνούμε ώστε οι απαιτήσει που απευθύνουμε σε δημόσιους θεσμούς ή συμβα... ιδιώτες να μην ε, μπερδεύονται. Γιατί μπορεί να οδηγηθούμε είτε σε διακρίσεις είτε σε στρεβλώσεις ακόμη και της αγοράς. Γι' αυτό και πιστεύω ότι ιδιώτες, εταίροι και δημόσιοι εταίροι θα πρέπει να εξετάζονται με την ίδια ε, προοπτική. Θα έλεγα ακόμα τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα έπρεπε να υπάγονται στους ίδιους κανόνες, για να το πω έτσι. Εν τέλει, βέβαια, δεν ξέρουμε εάν ο κανόνας των 30 ε, ημερών συνολικά ε, είναι σχεδιασμένο σωστά. Δηλαδή, πρέπει να κοιτάξουμε και να προστατεύσουμε τα συμφέροντα των μικροπιστών επιχειρήσεων, αλλά και του δημοσίου τα συμφέροντα. Και γι' αυτό μια μέγιστη ε, προθεσμία 60 ημερών, πιστεύω, είναι πιο λογική. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Σοντή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και εγώ θέλω να συγχαρώ τον εισηγητή και κυρίως για τον τρόπο με τον οποίο τονίζει το ρόλο των ΜΜΕ. Συμφωνώ απόλυτα στην ε, παρατήρηση ε, για την εφαρμογή των ε, και στις ευρωπαϊκές αρχές. Δηλαδή, δείτε και η Κομισιόν χρωστάει του κόσμου τα λεφτά στις, ε, στους διάφορους οργανισμούς ε, επιχειρηματολογώντας ότι δεν πληρώνει γιατί, γίνονται, γιατί γίνεται audit. Λοιπόν και θέλω εγώ να υποβάλω αυτή την, ε, αυτό το αίτημα στον εισηγητή γιατί δηλαδή και μεταξύ θεσμικών οργάνων, δημόσιων θεσμικών οργάνων όταν υπάρχουν πληρωμές και καθυστερημένες να μην εφαρμόζεται το μέτρο. Τώρα, επιστήνω την προσοχή σας ότι η εφορία θα φορολογεί αυτόματα. Ούτως ώστε η πρέπει... Πρέπει να λάβουμε μέτρα ούτω ώστε να εκπίπτουν από τη φορολογία όλοι οι τόκοι που επιφέρει το χρέος. Ο κύριος Κυλακάκης. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να τονίσω τη σχέση μεταξύ του δημοσίου κλάδου και των τοπικών αρχών. Οι τοπικές αρχές σε πολλές περιπτώσεις πληρώνονται από τον δημόσιο κλάδο, όχι όμως μέσω εμπορικών συναλλαγών. Και έχουν υποχρεώσεις έναντι των ιδιωτικών επιχειρήσεων πλέον τις οποίες δεν μπορούν, στις οποίες δεν μπορούν να ανταποκριθούν. Δεν μπορούν να προβούν σε πληρωμές μετρητής, γιατί ο δημόσιος κλάδος δεν τους ε, πληρώνει σε πολλά τμήματα, σε πολλές χώρες της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης και στη δική μου χώρα. Και ξέρω πώς λειτουργούν τα πράγματα, γιατί καθυστερούν οι πληρωμές από το δημόσιο κλάδο στις τοπικές αρχές. Και οι τοπικές αρχές αντιμετωπίζουν τεράστιες οικονομικές δυσκολίες σε ό,τι αφορά την πληρωμή μετρητής. Και ουσιαστικά τιμωρούνται για κάτι το οποίο, για το οποίο δεν ευθύνονται. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη λοιπόν αυτή τη σχέση μεταξύ των κρατικών φορέων και των τοπικών αρχών, ιδιαίτερα όπου μιλάμε για μεγάλα ποσά τα οποία διοχετεύονται στις τοπικές αρχές χωρίς οποιοδήποτε χρονικό πλαίσιο, οποιαδήποτε χρονική προθεσμία. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος, να δώσω στην κυρία Μπρίκμαν Μπρίκμαν το λόγο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και εγώ θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή. Οι τροπολογίες που προτείνει πάνε προς τη σωστή κατεύθυνση για τη βελτίωση της πρότασής μας ούτως ώστε να γίνει ακόμη πιο ευνοϊκή για τα συμφέροντα των ΜΜΕ που ξέρετε ότι αποτελούν και το βασικό αντικείμενο της αναθεώρησης οδηγίας τόσο για την τροπολογία, για τις ενημερωτικές εκστρατείες, για την, τον κώδικα συμπεριφοράς τον κώδικα αυτόματη εκτέλεση της πληρωμής των καθυστερημένων ε, πόσων και των τόκων κλπ. κλπ. Oh. Όλες αυτές οι τροπολογίες είναι πάρα πολύ επικοδομητικές και μπορούμε να συμφωνήσουμε σχετικά. Επιτρέψτε μου όμως να σταθώ σε ένα σημείο κλειδί μίας τροπολογίας που κατατέθηκε και ξέρετε ότι η Κομισιόν δεν συμμερίζεται την ανάλυση. Για τις ε, πληρωμές μεταξύ επιχειρήσεων, ξέρετε, Μίλησαμε για την ελευθερία σύνοψη ε, συμβάσεων κλπ. Δεν θα φλερίσω γι' αυτό, αλλά θέλω να είμαι σαφής. Υπάρχουν δύο διαφορετικές καταστάσεις, δύο διαφορετικά σενάρια σε περίπτωση εμπορικών συναλλαγών μεταξύ επιχειρήσεων έχουμε την περίπτωση όπου ΜΜΕ πραγματικά υποφέρουν από τεράστιες καθυστερήσεις πληρωμών που επιβάλλονται από μεγάλες επιχειρήσεις. Είναι κλασικές περιπτώσεις δηλαδή των επιχειρήσεων που ε, συνεργάζονται με μεγάλα δίκτυα διανομής ε, πρέπει να ε, λύσουμε σίγουρα αυτή την κατάσταση. Υπάρχει όμως και ένα άλλο σενάριο το οποίο πολύ συχνά ε, το ξεχνάμε. Οι ΜΜΕ πολύ συχνά ε, και αυτές ε, καθυστερούν να πληρώσουν. Έχουμε λοιπόν καθυστερήσεις πληρωμών μεταξύ χιλιάδων ΜΜΕ το να εναρμονίσουμε 60 μέρες για όλες τις περιπτώσεις και για όλους τους τομείς, όποια και να είναι η κατάσταση των ΜΜΕ, ε, δεν ε, θα είναι τόσο ευνοϊκό για αυτές τις ε, χιλιάδες ΜΜΕ που χρειάζονται αυτήν την ελευθερία. Λαμβάνοντας υπόψη λοιπόν αυτήν τη διαφορετικότητα των καταστάσεων, Θεωρήσαμε ότι μία τέτοια ενιοποίηση θα μπορούσε να, ε, να, βλα, να είναι επιβλαβής ε, για τις ε, ΜΜΕ και θα μπορούσε να, τις, να τους δημιουργήσει δυσχέρειες λαμβάνοντας υπόψη δηλαδή και την τωρινή κατάσταση ε, της κρίσης και της δυσκολίας πρόσβασης στα, στο δανεισμό είναι δύσκολο πράγμα Λοιπόν, αναζητούμε μια ισορροπημένη λύση. Ένας από τους σκεώδεις εισηγητές ζήτησε ότι πρέπει να, ζήτησε να βρούμε μια ισορροπημένη λύση. Και εμείς είμαστε υπέρ της ισορροπημένης λύσης, αλλά δεν πιστεύουμε ότι αυτή η ισορροπημένη λύση θα βρεθεί στο πλαίσιο της ε, ε, ενιοποίησης ε, της προθεσμίας πληρωμών για όλες τις επιχειρήσεις. και τα κράτη-μέλη το δέχτηκαν εκτός από ένα. Έχουμε λοιπόν εμείς πολλές εξαιρέσεις που πρέπει να τις διαχειριστούμε ανάλογα δηλαδή και με την ε, πολυπλοκότητα του τομέα. Δεν μπορούμε λοιπόν σε αυτό να συμφωνήσουμε με τον εισηγητή. Σας ευχαριστώ και επειδή έχει περάσει και ο χρόνος και δεν έχουμε διερμηνία στη διάθεσή μας ε, α, χωρίς περιορισμούς, θα ήθελα να σας ρωτήσω, θέλετε να κλείσουμε. Ευχαριστώ Πρόεδρε, εγώ θα είμαι πανσύντομος και γιατί μου φαίνεται ότι η συζήτηση πήγε πάρα πολύ καλά. Σχετικά δηλαδή με την πρώτη συζήτηση που είχαμε τον Δεκέμβριο έχουμε κάνει ένα σημαντικό βήμα προς τα μπρος. Εγώ μπορώ πλέον να πω ότι η κατεύθυνση είναι η σωστή. Αδιαμφισβήτητα πρέπει να εμβαθύνουμε ορισμένα θέματα. Και εγώ εξάλλου στην εισαγωγή μου για ορισμένα σημεία, για παράδειγμα η οροφή του 5% το business του business λέει ο μιλητής. Η σχέση μεγάλης επιχείρησης, μικρής επιχείρησης, πραγματικά νομίζω ότι για αυτά τα θέματα τάραξα τα νερά και μπορούμε να τα εμβαθύνουμε. Όπως επίσης και για όλη τη θεματική της σύναψη συμβάσεων, των συναλλαγών. Σημερίζομαι λοιπόν αυτή την παρατήρηση. Είναι ένα μέτρο το οποίο είναι υπέρ των ΜΜΕ διότι αποτελούν και το πιο σημαντικό και θεμελιώδες κομμάτι της ευρωπαϊκής οικονομίας. Εμείς λοιπόν θα πρέπει να προσανατολίσουμε αυτό το μέσο προς την υποστήριξη των ΜΜΕ. Η παλιά οδηγία δεν λειτουργήσε, αυτή η, λειτουργία, οδηγία πρέπει να λειτουργήσει. Με τα προβλήματα κρίσης που έχουμε, χωρίς δηλαδή δυνατότητα πρόσβαση στον δανεισμό, με την έλλειψη ρευστότητας κλπ. Άμα δεν λύσουμε αυτό το πρόβλημα, οι ΜΜΕ διατρέχουν να φαλυρίσουν και θα χάσουμε ένα σωρό λεφτά και θέσεις εργασίας και για το business του business που λέει ο μιλητής πρέπει να το προσέξουμε διότι αυτό το πρόβλημα πρέπει να το προσέξουμε και στις σχέσεις με τη μικρή επιχείρηση και με τη μεγάλη επιχείρηση είναι ένα σημείο το οποίο πρέπει να εμπαθύνουμε. πρέπει να βρούμε τη σωστή ισορροπία, τη σωστή σύνθεση <coughs> κρατώντας όμως τον μύτο της Αριάδνης για να μπορέσουμε δηλαδή να ενισχύσουμε την απασχόληση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξεπεράσαμε τις 12. Ευχαριστώ τους διερμηνείς. Ευχαριστώ πολύ. Thank you very much.